Euh, euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, οι πρόεδρος και όλοι οι αντιπρόεδροι απουσιάζουν. Οπότε εγώ η πρεσβυτέρα των φυλακών θα προεδρεύσω σε αυτή τη συνεδρίαση. Σας εύχομαι καλώς ήρθατε. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν παρατηρήσεις, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Θεωρείται εγκεκριμένη. Δεύτερο σημείο, η δημόσια κρόαση θα μιλήσω αγγλικά. Πρέπει να μιλήσω αγγλικά γιατί έχω τι σημειώσει μου αγγλικά. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τα αγγλικά μου. Δεν έχω ξφορδιανή προφορά όμω. Δημόσια ακρόαση όσον αφορά τι προοπτικέ να δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο Αποπληρωμή του Χρέου και να ε, θεσπιστούν ευρωμόλογα. Και η τελική έκθεση είναι η τελική παρουσίαση και σας καλωσορίζω. Σας κάλεσα στο Κοινοβούλιο να παρουσιάσετε την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο Αποπληρωμής του Χρέους και να εισαχθούν αυτά τα ομόλογα του ευρώ. Εκ μέρους της Επιτροπής σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων εργάστηκε τους τελευταιες 6 6-7 μήνες και εξέτασε τους κινδύνους, τις νομικές απαιτήσεις και τις ε, οικονομικές συνέπειες πρωτοβουλειών για αυτή την έκδοση αυτών των ευρωμολόγων που θα χρησιμεύσουν τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αποπληρωμής του Χρέους Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμεύσε πολύ, ζήτησε να συσταθεί αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων και είμαστε ικανοποιημένοι ε, που είσαστε εδώ για να παρουσιάσετε τα πορίσματά σας. Λάβαμε την τελική σας έκθεση πριν από μερικές ώρες, οπότε όπως τα καταλάβατε δεν είχαμε το χρόνο να διαβάσουμε με όλες τις λεπτομέρειες το κείμενο, ακόμα δεν είχαμε το χρόνο και γι' αυτό προσβλέπουμε στα σχόλιά σας. Ε, οι εισαγωγικές παρατηρήσεις θα γίνουν από την κυρία Τούμπελ Γκιούγκερελ που είναι πρόεδρος της ομάδας εμπρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας καλωσορίζουμε, σας γνωρίζουμε βέβαια από το παρελθόν σας στη θέση σας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, και έχετε ένα δεκάλεπτο για να παρουσιάσετε την έκθεση. Ε, μετά θα ακολουθήσουν διάφορες δηλώσεις από πλευρά των μελών της ομάδας εμπειρογνωμόνων που είναι ε, παρόντα. Θα κάνω τη σύσταση όταν θα πάρουν το λόγο και θα έχουν ένα 7 λεπτό στη διάθεσή τους ο καθένας και δίνω το λόγο αμέσως στην κυρία Τρούμπελ Γκούγκελχελ. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της ε, Επιτροπής, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσω τα πορίσματα της εκθεσής μου σήμερα μαζί με τους συναδέλφους, τέσσερα από τα μέλη της ε, Επιτροπής και θα ήθελα σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας για να προωθηθεί το όλο θέμα. Πάνω από δύο χρόνια πριν έγιναν δύο προτάσεις σχετικά με το θέμα αυτό και αν θυμόσαστε ποια ήταν η κατάσταση πριν από διετία μπορείτε να δείτε την έκθεσή μας και να δείτε το παράρτημα που τη βλέπετε σελίδες 2 και 6 και 4 τα spreads των διαφόρων κρατικών ομολόγων που έπρεπε τότε να καταβάλλονται. Πολύ ψηλά επιτόκια. Εν τω μεταξύ η κατάσταση άλλαξε, έγιναν μεταρρυθμίσεις από τις διάφορες ε, κυβερνήσεις. Ε, πρόσφατα ε, προωθήθηκε, θεσπίστηκε η Τραπεζική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δραστηριοποιήθηκε. Μπορεί να διαρωτηθείτε, υπάρχει ακόμα ανάγκη για δράση. Αυτό εξαρτάται από τη δική σας αξιολόγηση όσον αφορά το μέλλον της Ένωσης και την μορφή που θέλετε να έχει αυτό το μέλλον. Η πρώτη ιδέα παρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια, δημιουργία αυτού του Ταμείου Πληρωμή του Χρέου και να συναυθεί ένα σύμφωνο για την απληρωμή του χρέου και ύπαρξη κρατικού χρέου πάνω από 60% του ΑΕΠ θα μεταφερόταν σε ένα κοινό ταμείο αυτό θα μείωνε τα επιτόκια για τι χώρε που είχαν υψηλότερο χρέο και θα επέτρεψε στις χώρε αυτέ να μειώσουν το υπερβολικό του χρέο. Σε αντάλλαγμα, οι κυβερνήσει θα έπρεπε να, κάνουν, να αναλάβουν δεσμεύσει για εξυγίανση των δημοσιονομικών για τη διάρκεια, διάρκεια ζωής του Ταμείου. Δεύτερη ιδέα που επίση συζητείται αρκετά χρόνια είναι η ιδέα των ευρωομολόγων και αυτό θα προέβλεπε κοινή έκδοση βραχυπρόθεσμων τέτοιων κρατικών ομολόγων το DRF, αυτό το ταμείο, θέλει να αποκαταστήσει τα δημοσιονομικά αφαιρώντας το κίνδυνο ε, του χρέους όταν οριμάζει το χρέος και να δημιουργηθεί ποικιλοποιημένο ενεργητικό, σε ρευστό και να ολοκληρώσει την ενοποίηση τη αγορέ και να εξηγιανθεί η αγορά και τελικά να μειωθεί το υπερβολικό χρέο στην Ευρωζώνη. Η ιδέα των ευρωμολόγων εστιάζεται σε διαφορετικό στόχο, έχει σαν στόχο τη σταθεροποίηση των αγορών χρέου των κυβερνήσεων, αφαιρώντα τον κίνδυνο ε, μετακύληση του χρέου και για να υπάρχει καλύτερη ενοποίηση των χρηματοσυντικών αγορών μέσω τη δημιουργία ενό βραχυπρόθεσμου ε, στοιχείου ενεργητικού σε μετρητά και η νομισματική πολιτική θα έπρεπε να στηρίζεται και να διαδίδεται. Ε, περίπου 1,8 με 3,1 τρισεκατομμύριο ε, ευρώ χρέους θα πήγαιναν στο ταμείο και θα πήγαινε το μέγιστο μέγεθος του πόρου από 1,7 στα 2,85 ε, τρισεκατομμύρια. Θα πρέπει να αναλάβουν υποχρεώσεις τα κράτη-μέλη για τη διάρκεια ζωής του Ταμείου που θα είναι 10 με 25 χρόνια. Κανείς θα μπορούσε να επιλέξει ένα ταμείο που θα ε, περιέχει διάφορες εγγύσεις και αυτό χρειάζεται τεράστιες δεσμεύσεις και συνεπάγεται αλλαγή ε, των συνθήκων. Ε, μια καταναλογία, εγγύσεις καταναλογία δεν θα πετύχανε το σωστό επί της οικονομίας σε τόκους. Ποιος είναι ο κίνδυνος. Θα ωφελούνται απε, απευθείας οι χώρες και θα έπρεπε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους σε μακρά χρονική περίοδο. Οι κίνδυνοι που διαβλέπονται είναι η έλλειψη της ευελιξίας και αύξηση των επιτοκίων για χώρες με υψηλή βαθμολόγηση όσον αφορά τη χρηματοστητική δυνατότητα. Ε, και οι βασικοί κανόνε για δημοσιονομική πολιτική εκ των προτέρων από πολύ πριν θα πρέπει να καθορίζονται και θα πρέπει να είναι δύσκολο να υπάρξει συμμόρφωση σε τη διάρκεια τη χρονική. Η ομάδα διερεύνησε εναλλακτικέ λύσει, ένα μικρότερο ταμείο με ίσο μερίδιο του χρέου όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ από κάθε χώρα και, και συντομότερη διάρκεια ζωή του ταμείου. Αυτή η μεταβλητή θα έχει ωφέλη και θα μειώνει σε κάποιο βαθμό του κινδύνου. Αλλά δεν θα επέλυε το πρόβλημα διαφοροποιημένων επιπέδων ε, χρεών από, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα ευρωμόλογα θα μπορούσαν να έχουν κοινή ε, Κοινέ εγγύσει ή αναλογικέ εγγύσει το μέγεθο του ταμείου θα εξαρτάται από, τις από τα ποσά που καλύπτονται και αν συμπεριλαμβάνονται αξιόγραφα μέχρι δύο έτη, αναμένεται ότι το μέγεθο θα είναι περίπου 0,8 δισεκατομμύρια βάσει των στοιχείων για τα εφιστάμενα χρέη, τα βραχυπρόθεσμα και το μέγιστο μέγεθο του ταμείου, εάν το όριο 30% κρατικού χρέους διατηρηθεί, θα μπορούσε να είναι σαν ταμείο στα 1,8 δισεκατομμύρια. Ένα χρέο κάτω από ένα χρόνο σημαίνει ένα ταμείο που ένα αναμενόμενο ποσό περίπου 0,5 τρισεκατομμύριο και μέγιστο μέγεθο θα μπορούσε να είναι 0,9 τρισεκατομμύρια αν το λογικό όριο καθοριστεί για το χρέο που θα είναι 10% του ΑΕΠ. Τα ευρωμόλογα με κοινέ και πολλέ εγγυήσει θα μπορούσαν να απαιτούν τροποποίηση των συνθεκών. Με αναλογικέ εγγυήσει αυτό μπορεί να μην μπορεί να γίνει οι χρηματοδοτιστικές συνέπειες θα είναι ακόμα μικρότερες και ο αντίκτυπο πρωταρχικά θα ήταν ποιοτικού είδου. Η δημιουργία ενός προσωρινού ταμείου συζητήθηκε, αλλά στην πράξη θα ήταν δύσκολο να διαλυθεί ένα τέτοιο ταμείο από τη στιγμή που θα ιδρυόταν. Ένας από τους κινδύνους των ευρωμολόγων θα ήταν ότι μπορεί να οδηγήσει σε υπερεξάρτηση όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο χρέος. Πέρα από τους οικονομικούς σωματοστικούς κινδύνους που ήδη ανέφερα, τώρα σε εξηγήσω τι έχουμε, αυτό που περιγράψαμε σαν ηθικό κίνδυνο, δεντρολογικό κίνδυνο και συνάδελφοι θα εξηγήσουν τις λεπτομέρειες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ηθικός κίνδυνος είναι εκείνοι που μπορεί να εκμεταλλευτούν το όλο σύστημα. Σημαίνει ότι μια χώρα αναβάνει τον κίνδυνο και άλλη χώρα, η άλλη ομάδα χωρών ε, πληρώνει το κόστος από τη στιγμή που πραγματοποιηθούν και υλοποιηθούν οι κίνδυνοι. Τι μπορεί να γίνει όσον αφορά αυτό το κίνδυνο, τον διοντολογικό. Συζητήσαμε τέσσερι δυνατότητε, παραδείγματο χάρη, δεσμευτικέ υποχρεώσει, συμπληρωματικέ εξουσίε παρεμβάσεω για εκείνου που διαμορφώνουν ευρωπαϊκή πολιτική σε περίπτωση μονή, σε μη συμμόρφωση με συμπεφωνημένε πολιτικέ, κίνητρα οικονομικά και απειλή αποκλεισμού από, από μηχανισμούς κοινή έκδοσης που συζητούνται στην ομάδα. Τώρα θα ήθελα κροθυγώς να αναφερθώ στις νομικές απαιτήσεις όταν συζητάμε αυτά τα συστήματα για την έκδοση των ομολόγων. Οι συνθήκες οι παρούσες δεν επιτρέπουν την κοινή έκδοση με κοινέ και αρκετές εγγύσεις μπορεί να επιτρέπουν αναλογικά συστήματα όπω κεφαλαϊκέ δομέ, αναλογία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίηση. Οι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνουν αρκετέ αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουν ένα τέτοιο ταμείο αποπληρωμή του χρέου ή να εκδώσουν ευρωμόλογα μέσω τη νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Το να δοθούν χρηματοστικέ αρμοδιότητε είναι σαν να δώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξουσίε να θέσουν ανησυχίε όσον αφορά εθνικού προπολογισμού και απαιτούνται αλλαγέ των συνθήκων. Κάποια εθνικά συνταγματικά δίκαια απαιτούν όρια όσον αφορά τι εθνικέ ευθύνε και να τίθενται εκ των προτέρων και τακτικέ ψηφοφορίε πρέπει να λαμβάνουν χώρα όσον αφορά πρόσθετε υποχρεώσει. Όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμότητα, σίγουρα θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί η κοινοτική μέθοδο σε περίπτωση που διάφοροι μηχανισμοί για την κοινή έκδοση δημιουργηθούν. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχο θα πρέπει να προβλέπεται με έναν τρόπο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώ και τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν ε, ε, λόγο στην λειτουργία οποιοδήποτε μέσου για την κοινή έκδοση. Η έκθεση, έκδοση συγγνώμη. Και η έκθεση τονίζει επίση ότι οι μηχανισμοί κοινών εκδόσεων δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τι προσπάθειε που καταβάλλονται από τα κράτη-μέλη για να μειώσουν τα χρέη του και να κάνουν πολιτικέ, να εφαρμόσουν πολιτικέ ε, μεταρρυθμίσεων. Κλείνοντα, η κοινή έκδοση θα έχει ωφέλη γιατί θα σταθεροποιούσε τι αγορέ χρεών των κυβερνήσεων, στηρίζοντα νομισματική πολιτική τη μετάδοση αυτή και οδηγώντα σε χρηματοστατική σταθερότητα και την ολοκλήρωση, οικονομική και χρηματοστατική κίνδυνη και ηθική κίνδυνη και αυτοί πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό ίσως να θεωρηθεί συνετό πρώτα να συλλεχθεί εμπειρία με την μεταρρυθμισμένη οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης πριν ληφθεί αδίποτε απόφαση για μηχανισμούς κοινής έκδοσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Κυρία Τούπερ Γκούγκερελ, είναι φρόζεκτες γιατί μόλις λάβαμε το κείμενο της εκθέσεως. Τώρα λοιπόν ακούμε τα λοιπά μέλη της ομάδας επιρρογνωμόνων. Η κυρία Άνια Κερασί Μπενή, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Παρισιού, καθηγήτρια οικονομικών και πρόεδρο του Γαλλικού Συμβουλίου Οικονομικών Αναλύσεων. Κύριε Μπένασή, κύριε, έχετε το λόγο. 7 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά για να διατηρήσουμε κοινή γλώσσα με τους τρεις συναδέλφους. Μου ζητήθηκε να παρουσιάσω τους στόχους ε, της έκδοσης των ε, ευρωομολόγων. Ξέρετε, ο αρχικός στόχος του Ταμείου Αποπληρωμής και του Σχετικού Συμφώνου και του Ευρωομολόγου οι στόχοι των δύο ήταν διαφορετικοί αρχικά για το σύμφωνο για την αποπληρωμή του χρέους. Ο στόχος ήταν η γεφύρωση των προβλημάτων ε, και ο περιορισμός των δημοσιονομικών δαπανών ή του κόστους για τις χώρες αυτές, ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης του χρέους. Ενώ για το ευρωομολόγο στόχος ήταν να αντιμετωπιστούν κρίσεις ρευστότητας και να ενισχυθεί η δημοσιονομική σταθερότητα και μια οικονομική διαχείριση χωρίς προβλήματα. Τώρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε τρεις διαφορετικούς στόχους. Μπορούμε να πούμε ότι ενισχύουμε την βιωσιμότητα του χρέους, ενισχύουμε την σταθερότητα στις αγορές του χρέους και συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην οικονομική επανένταξη και σταθεροποίηση. Θα σχολιάσω λοιπόν τους τρεις αυτούς στόχους. Πρώτα την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους μέσω του περιορισμού του κόστους χρηματοδότησης σε χρονικά όρια φυσιολογικά. Και εδώ θα πω ότι και για τις χώρες με χαμηλό χρέος είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για όλους φυσικά, να μπορούν οι χώρες με μεγάλο χρέος να περιορίζουν το κόστος του δανεισμού διότι έτσι χρειάζεται να εξασφαλίσουν πρωτογενές πλεόνασμα πολύ, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι χώρες αυτές με τρεις κινδύνους. Πρώτον το, το επίπεδο της ανάπτυξης, τον πολιτικό κίνδυνο βεβαίω και τον κίνδυνο τα κυβερνήσει των κρατών αυτών να μην έχουν επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια για να κάνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μεγάλου ελληνικού. Έτσι λοιπόν ε, είναι απαραίτητο να μην είναι υπερβολικά υψηλό το κόστος του δανεισμού για κανέναν. Ε, δεύτερον, σε ενοποιημένου όρου, η δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίστοιχη με αυτή των ΗΠΑ. Πολύ καλύτερη από αυτή τη Ιαπωνία. Ο μόνο λόγο λοιπόν για τον οποίο το ε, κρατικό χρέο μπορεί να έχει περισσότερου κινδύνου από ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου είναι η απουσία αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και οι ανισορροπίες μεταξύ των ε, κρατικών και των νομισματικών ορίων. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος της αναχρηματοδότησης και να βοηθήσουμε τα κράτη να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Οι επιπτώσεις μιας κοινή έκδοσης για την αναχρηματοδότηση του κόστους, για για τον επιμερισμό δηλαδή του κόστους της χρηματοδότησης, μπορεί να μην φαίνεται ε, εκ πρώτης όψεως, γιατί το κόστος μπορεί να θεωρείται ότι θα προκύψει εάν εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ε, φερεγγιότητα από το κοινό σύστημα έκδοσης και εάν το κέρδος από την ρευστότητα, στην περίπτωση της κοινή έκδοσης, μπορεί να ξεπεράσει την απώλεια ρευστότητας από το εθνικό χρέος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι δυνατόν ε, να περιοριστεί το συνολικό κόστος του κρατικού χρέους, χωρίς όμως αυτό να είναι δεδομένο εάν δεν υπάρξει ενισχυμένη φερεγγιότητα ε, όλες τις προσπάθειες αυτές Θα περάσω τώρα στο δεύτερο στόχο, που είναι η ενίσχυση της σταθερότητας στην αγορά του χρέους και η μείωση του κόστους ε, χρηματοδότησης αναχρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα υψηλό επίπεδο χρέους, το οποίο με τη ισχύοντα πάντα θα είναι εκτεθειμένος σε κρίσεις με σημαντικές επιπτώσεις και μεταξύ κρατών μελών αλλά και ε, σε επίπεδο δανεισμού μεταξύ κρατών και από κράτη σε τράπεζες ή από τράπεζες σε κράτη καλύτερα. Ένα στόχος λοιπόν θα ήταν να περιοριστεί το πεδίο, η απο σε κρατη καλυτερα ενα στοχος λοιπον θα αυτού του κινδύνου ρευστότητας και να αποτραπεί να αποτραπούν δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά, αλλά και να ρυθμιστούν κάποια προβλήματα συμπεριφοράς στους επενδυτές. Αντίστοιχα θα είχαμε λιγότερη αρνητική, λιγότερο αρνητικό αντίκτυπο ε, κυκλικό για τις ε, τράπεζες αλλά και για το κρατικό χρέος. Και έτσι θα βελτιωνόταν οι δυνατότητε χρηματοδότηση από πλευρά των τραπεζών, φερειπίν για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτό θα σήμαινε καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και χαμηλότερα επίπεδα δανεισμού, επιτόκια δανεισμού δηλαδή, ακόμη και σε περιπτώσεις κρίσεω. Μπορούμε έτσι να περιμένουμε μία πιο ασφαλή πρόσβαση στην αγορά, ακόμη και σε περίπτωση ασυμμετρικών μακροοικονομικών κλειδονισμών και αποκατάσταση ε, του επιμερισμού του κινδύνου μακροοικονομικά. Τώρα θα ήθελα να περάσω ε, στον, άλλο, στον τρίτο στόχο που είναι να συμβάλλουμε στην επανένταξη και τη σταθερότητα σε οικονομικό επίπεδο πάντα. Οι τράπεζες λοιπόν στην Ευρωζώνη χρειάζονται ενεργητικό που μπορεί να αξιοποιηθεί ως ε, ε, εξασφάλιση ρευστότητας ή μπορεί να απολυθεί σε σχετικά σταθερές τιμές ή να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για διαδικασίες επαναχρηματοδότησης. Η ύπαρξη τέτοιου είδους ενεργητικού στη ζώνη του ευρώ θα μειώσει, θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις από την ε, επιδίνωση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας για τα επιμέρους κράτη-μέλη στο... και τη δυνατότητα για πρόσβαση ε, στη χρηματοδότηση. Θα μπορούσαν δηλαδή τα κοινά αυτά ενεργητικά, επιμεριζόμενα ή αναπτυσσόμενα από κοινού να αποτελέσουν μια πολύ καλή εγγύηση και να μειώσουν την εξάρτηση από την αξιολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας του κράτους για τις τράπεζες και τις ε, επιχειρήσεις. Επίσης, μπορούμε να περιμένουμε μείωση του κινδύνου αποσταθεροποίησης σε περιπτώσεις κρίσεως. Και κλείνοντας, θα θέλω να πω ότι μπορεί να μην υπάρχει συνένεση μεταξύ των εμπειρογνωμών ω προ τι συνέπειε μια κοινή έκδοση αλλά και τι συμφωνούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του κατακαιρματισμού της αγοράς, οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν, διαφωνούν καλύτερα ως προς την έκταση της επιπλέον ε, βοήθειας και στήριξη που μπορεί να προσφέρει το σύστημα αυτό της κοινή έκδοσης. Πιστεύω λοιπόν ότι από τους τρεις στόχους που αναφέρουμε ίσως δεν μπορέσουν να επιτευχθούν και οι τρεις με το σύστημα αυτό, το σύμφωνο δηλαδή κοινή έκδοση και το ευρωομολόγο, γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια επιλογή με προτεραιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμών είναι η Μπεατρίς Βιτάλντι Μαουρό που είναι καθηγήτρια στο, ε, στο Πανεπιστήμιο για μακροοικονομικά, για θέματα μακροοικονομικών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα μιλήσω αγγλικά και θα ήθελα να αρχίσω με το όλο ιστορικό αυτού του ε, Ταμείου Αποπληρωμής ή Απόσβεσης όταν ε, τα ε, μέλη του Γερμανικού Συμβουλίου ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, ε, αντιμετωπίσαμε πολλές αντιδράσεις, δηλαδή πλήρη απόρριψη από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά αποδοχή άλλων μερών της πρότασης. Αισθανθήκαμε όμως ότι δεν υπήρχε κατανόηση του συνολικού πακέτου γιατί έτσι θα έπρεπε να θεωρηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για τα βασικά συστατικά ε, αυτού του πακέτου. Ένας μηχανισμός αντιμετώπισης της ε, κρίσης όπου μέσω της ε, κοινή έκδοσης θα αποσβέσει τους κινδύνους επαναφοράς. Επίσης, να αντιμετωπίσουμε το συνολικό θέμα του χρέους ε, μέσω backloading αυτής της ε, διαδικασίας και επίσης να ανταποκριθούμε στις χώρες που έχουν ενταχθεί στο ε, σύμφωνο σταθερότητας και είναι αξιόπιστα για αυτές τις δεσμεύσεις μέσω ε, ενός ε, premium αξιοπιστίας και μετά να δούμε υπό ποιους όρους μπορεί να ισχύσει ένα σχήμα μη διάσωσης μέσω ενός ταμείου απόσβεσης ε, του χρέους. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι λαμβάνουμε υπόψη ένα μακροχρόνιο καθεστώς για να φτάσουμε εκεί που διαφέρει από το παρόν, διότι μιλάμε για κοινή έκδοση όπου θα υπάρχει αμοιβεοποίηση του χρέους, αλλά περιορισμένη στην ε, ε, αμοιβεοποίηση που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Άρα Αυτό που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίσουμε το χρέος και την διαιώνισή του. Ε, αν θέλετε μία εικόνα, σκεφτείτε το ταμείο ως ένα βουνό με πολλές, με υπόρειες που συνεχίζουν μέχρι το επίπεδο της θάλασσας. Ενώ τα κοινά προγράμματα έκδοσης ε, έχουν μία ε, είσοδο και στη συνέχεια μία διάρθρωση που όλο ένα και διονγκούται. Το σχήμα λοιπόν για το Ταμείο Απόσβεσης Χρέους ε, εξετάζεται ιδιαίτερα στο έγγραφο που σας έχω δώσει. Καταρχήν υπάρχει η αρχική πρόταση που περιλαμβάνει ένα μεγάλο βουνό, ας το πω έτσι, διότι αμοιβεοποιεί όλο το χρέος που ανέρχεται πάνω από το 60% του ΑΕΠ. Άρα στο υψηλότερο σημείο θα είχαμε μια κοινή έκθεση της τάξης των 2,83 ευρώ. Αυτό το συζητήσαμε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κατόφλι από 60 σε υψηλότερο αριθμό, δηλαδή ε, αναφέρεται και το 75% του ΑΕΠ. Υπάρχουν όμως οι χώρες που θα ευεργετηθούν περισσότερο από αυτό το ταμείο σε σχέση με άλλες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες γιατί έχουν υψηλότερο ε, χρέος. Ε, θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε ένα πιο ισοβαρές σχέδιο, δηλαδή κάθε χώρα να συμμετέχει ε, σε μία τάξη του 20% του ΑΕΠ. Σε αυτή την τάξη μεγέθους έτσι θα υπάρχει ένα διαφορετικό μερίδιο και θα υπήρχε συγκρισιμότητα και στην έκδοση ευρωομολόγων. Και το ανώτατο σημείο θα ήταν 1,73. Εάν μόνο το 20% αμοιβεοποιηθεί, το 20% του ΑΕΠ. Αυτό αυτό όμως ε, δεν θα οδηγήσει στην απαλυφή του χρέους για όλες τις χώρες. Ως προς τις εγγυήσεις ε, υπάρχουν διάφορα σχήματα εγγυήσεων και αυτό έχει πολλά πλέον εκτήματα αλλά και κινδύνους. Γι' αυτό χρειάζονται δικλίδες ασφαλείας. Μιλήσαμε για ένα καταναλογία σχέδιο όπου χρειάζονται άλλες ρήτρες ασφαλείας, δηλαδή σε ένα καταναλογία ε, σύστημα χρειάζεται, χρειάζονται κεφαλαιακές εισρωές. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζονται πολλές ε, ρήτρε, ε, καταρχήν δεσμεύσεις, το μέσο των δεσμεύσεων, όπως ορίζεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας, και να δούμε τι θα συμβεί για όσους δεν συμμορφούνται ε, σε αυτή την ανάβαση του βουνού και στη καθοδική πορεία θα είχαμε τα mark-ups στο σύστημα επιτοκίων, καθώς και άλλους μηχανισμούς που συζητήθηκαν στην έκθεση για να υπάρξει συμμόρφωση με τη μείωση του επίπεδου χρέους. Επίσης υπάρχει και το σχέδιο αναμόρφωσης όπου υπήρχε ένα κατόφλι χρέους που θα όριζε το επίπεδο δανειοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, δηλαδή να έχουμε ένα κατόφλι ως ε, παράγοντα σταθερότητας. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες ε, ασχολήθηκαν με αυτό το καθεστώς ε, αναδιάρθρωσης. Πολλοί εμπειρογνώμονες θεώρησαν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο διάσωσης σε αυτή την περίπτωση και μακροχρόνια θα πρέπει να εισαχθεί αυτός ο μηχανισμός, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός που θα υπερέχει των εθνικών ε, προϋπολογισμών. Αυτό σημαίνει αλλαγές στις συνθήκες. Όπως ανέφερε και η Πρόεδρος, εδώ υπάρχουν και νομική, νομικές επιπτώσεις, γι' αυτό χρειάζονται ε, αλλαγές στις συνθήκες αλλά σε μια διακυβερνητική διάρθρωση θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλους τύπους προτάσεων που έχουν ήδη εισαχθεί στην πρόταση που έχετε ενώπιον σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βεντάλντι Μάουρο. Τώρα είμαστε στην ισότητα των φίλων και περνάμε σε άρενα στον κύριο Γκαμπίσοφ που είναι σύμβουλος και εμπειρογνώμων για οικονομικά θέματα και χρηματοστατικά θέματα ευρωπαϊκά. Κύριε Μπίσοπ, έχετε το λόγο για ένα 7 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Περίπου πριν από δύο χρόνια, μια ομάδα εργασία από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Οικονομική Συνεργασία, ο Βουν και ο Βουν ήταν πρόεδρο, δημιούργησε το σχέδιο αυτό για τα ευρωμόλογα και διάφορε δομέ για εγγύσει. Όμω για λόγου νομικού που αναφέρθηκαν επακριβώ στην έκθεσή μα, κατέληξα στην άποψη ότι μόνο μια καταναλογία εγγύηση θα ήταν πολιτικά και νομικά εφικτή γι' αυτό παρουσιάσα τη δική μου μεταβλητή ένα σχέδιο για προσωρινό ταμείο για τα ευρωμόλογα TEF στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Βεβαίω, οι συμμετέχοντε στην αγορά έχουν απόψει για τι διευθετήσει που του ικανοποιούν. Όμω τα κοινοβούλια θα πρέπει και σωστά να προστατεύσουν μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα των εκλογίων του. Λοιπόν, ε, η η τέχνη ποια είναι, να βρούμε τη μέση οδό και αυτό που θα προσπαθήσω να συζητήσω βάσει της αναλύσεως της ομάδος. οικονομικέ οικονομικές πτυχές. Καταρχάς μόνο οι χώρες Ευρωζώνης που είναι σε καλή θέση στο Ευρωγκρουπ μπορούν να δανειστούν και αυτό ενισχύει την, το υπεστάμενο ε, πλαίσιο διακυβέρνησης. Λοιπόν, από δύο χρόνια ορίμανση, εν μία νυχτή θα μπορούσαν να περάσουν θα, θα περάσουν στα πέντε χρόνια για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να έχουμε μια δοκιμαστική περίοδο, ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν να εξετάσουν κατά πόσο ο μηχανισμό θα είναι μόνιμο, αν είναι επιτυχή και μόνο. Βέβαια, η έκδοση θα μπορούσε να σταματήσει από εκείνου που παίρνουν αποφάσει οποιαδήποτε στιγμή. Μετά θα πρέπει να σκεφτούμε τα εθνικά κοινοβούλια που θα πρέπει να έχουν τον οικονομικό έλεγχο, δημοσιονομικό έλεγχο και να ανανεώνουν το ταμείο κάθε πενταετία, Φερρυπίν. Όλοι στι συμμετέχουσε χώρε θα απαγορεύεται να μπορούν να αντλήσουν πόρους ε, κάτω από δύο χρόνια εκτός αυτού του TEF. Οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν τότε να μετακυλήσουν ε, τα ρημάζοντα ομόλογα δανειζόμενα από το TEF ανάλογα με την έκθεσή τους. Και αυτό αφαιρεί, αφαιρεί το κίνδυνο μετακύλησης και αυτό είναι κάτι που συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα. Θα υπάρχουν εξουσίες για το Ταμείο, το TEF, να μπορεί να αγοράζει ομόλογα όταν η ζωή των εφισταμένων ομολόγων είναι κάτω από δύο χρόνια. Οπότε το μέγεθος είναι κατά ελάχιστον 0,8 τρισεκατομμύρια, πιθανότατα 0,9-1,2 τρισεκατομμύρια και για κάτι σαν Ευρωπαϊκό Ταμείο που θα μπορούσε να γίνει αυτό θα έχουμε το μέγιστο 1,8-1,9 τρισεκατομμύρια. Βέβαια σημειώστε ότι το μέγεθος είναι θέμα πολιτικής επιλογής από τους λαμβάνοντες αποφάσεις στην Ευρώπη να διευρύνουν ή να συρρυκνώσουν το μέγεθος ανάλογα με θέματα της αγοράς και τα θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Χειριζόμενοι το, τον ηθικό κίνδυνο. Έχουμε τα ευρωμόλαγα, Ήδη έχουμε ε, τέτοιους κινδύνους. Ποιες είναι οι νομικές πτυχές. Το ETF μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρί να αλλάξει η συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιοδήποτε μηχανισμό για να απαγορεύσει κάποιου από του συμμετέχοντε να έχουν οικονομιστική κυριαρχία θα μπορούσε να είναι εκτός ε, των δικαιοδοσιών που προβλέπει η συνθήκη. Αυτή η δικασία λήψη αποφάσεων για αυτή την κοινή κυριαρχία θα απαιτεί διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ των συμμετοχών των κρατών και αυτό μπορεί να εδράζεται επί του μοντέλου για την ε, οικονομική νομισματική σταθερότητα στο σταθεροποιητικό μηχανισμό. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια τεχνική δομή για την έκδοση των ομολόγων βάσει του κανονισμού, βάσει του άρθρου 352 των συνθήκων. Και αν η συνθήκη ξανααναλυθεί και ξανασυζητηθεί σε μελλοντική, σε μελλοντική φάση και να υπάρξει κάποιο σύμφωνο με το στοτικό, τότε μπορούμε να φέρουμε ένα τέτοιο ταμείο TEF μέσα στο όλο πλαίσιο, αφού θα αναθεωρηθεί η συνθήκη. Οι μηχανισμοί τώρα, ποιοι είναι ο μηχανισμός. Ε, πρέπει να είμαστε απλοί ε, χρηματοδότης αγοράς που θα πρέπει να αντίθεται συμμετέχοντα κάτι μέλα. Λοιπόν, τα λεφτά που μπαίνουν εξισούνται με αυτά που βγαίνουν. Λοιπόν, η δομή για τη λήψη αποφάσεων είναι οι Υπουργοί Οικονομικών που αποφασίζουν και είναι υπόλογοι στα εθνικά του κοινοβούλια. Η δομή του κεφαλαίου, μέτριο ε, κεφάλαιο ε, και ελεγχόμενο και κανόνε και όρια για να αποφεύγεται τα μέλη να μειώνουν υπερβολικά το στάδιο ρημότητα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε ένα όριο. μέσω όρου του χρέου θα πρέπει να είναι πάνω από 7 χρόνια και κάτι κρίσιμο θα πρέπει να είναι ένα μέγιστο ποσοστό χρέου κάτω από δύο χρόνια, που έχει διάρκεια ζωή κάτω από δύο χρόνια. Ένα στόχο περίπου 25% και ένα όριο περίπου 35%-30%. Αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει να επανακαθοριστούν ίσω λεπτομερώ. Αποκλεισμό, εξαίρεση, είναι ε, κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Αν μια χώρα υπόκειται σε κυρώσει, τότε θα πρέπει να εξαιρείται. Δεν έχει νόημα να εγγυείται κανείς ένα κράτος το οποίο δεν είναι βιώσιμο το κρατικό χρέος. Και αυτό ε, πηγαίνει παράλληλα με μια πρόσκληση εντός εισαγωγικών μια χώρα να, να αναλάβει ένα πρόγραμμα του μηχανισμού σταθεροποίησης. Άρα ο ρόλος του εγγυητού δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την ευθύνη του έναντι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης. Θα πρέπει ε, να πηγαίνουν και σε ιδρύματα και σε άτομα ίσως αυτά τα ομόλογα. Ποια είναι τα ενδεχόμενα αποτελέσματα θα έχουμε ενεργητικό πάρα πολύ ρευστό, θα μειώσουμε το φαύλο κύκλο μεταξύ τραπεζών και κρατικού χρέους ε, τουλάχιστον κατά ένα τρίτο και εξαρτάται πώς θα γίνει τουλάχιστον θα πρέπει να θα χάσουμε το ένα τρίτο του χρέους. Θα βελτιώσουμε λοιπόν και την ποιότητα των τραπεζών σε αφορά την ε, ε, πιστοληπτική ικανότητα και θα μπορούμε να εφαρμόζουμε πιο ομαλά την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ευρωζώνη. Και τα ομόλογα του TF θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες και τους ασφαλιστές. Οι παρόντες κανονισμοί αφήνουν τα χρηματοστικά ιδρύματα πολύ λίγες αναλλακτικές, απλώς τα, εθνικά ομόλογα να τα μετακυλούν σε ομόλογα TF, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Πιστεύω θα υπάρχει ζήτηση στην αγορά. Κλείνοντας λοιπόν, έχουμε ενδεχόμενα, ας πούμε το χρυσό σενάριο πρώτα απ' όλα, Μ' αρέσει πάντα αυτό να ξεκινά από το καλό του χρόνου το 2015 με την εμπειρία του 5ου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που φαίνεται καλό και το Tupac να λειτουργεί καλά στο δεύτερο γύρο αυτού, θα έλεγα ότι αυτό θα μας έδινε μια καλή βάση όσον αφορά την εμπειρία να δούμε και να ξεκινήσουμε το TEF, αρχικά ξεκινώντας με το ελάχιστο μέγεθος αυτού. Το 2016 έχουμε λοιπόν, όσο γίνεται η και λοιπά και μετά τα χρόνια, οι, οι αρμόδιοι αποφασίζουν να επεκτείνουν ε, το ταμείο αυτό με αιτήσιε αποφάσει ανάλογα με την εμπειρία του κάθε εξαμήνου ξεκινώντας ε, με ένα ομόλογο που έχει οριμότητα 6 μήνε και ίσω μέχρι το 2018 αυτό το όριο να προχωρήσει σε 2 χρόνια πιο πέρα, πιο κάτω. Και σε αυτή τη φάση θα πρέπει να δούμε ένα μέγεθο που είπα που θα φτάνει περίπου τα 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι de facto ένα ευρωπαϊκό ταμείο σε αυτό το ύψο και τότε το TF, το ταμείο θα είναι 50% μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο φορέα και προφανώς αυτά τα ομόλογα θα είναι στοιχείο ενεργητικού για ποσοτική μίσθωση αν κάτι τέτοιο ε, θεωρηθεί ενδεικνυόμενο. Και ποιο είναι το μαύρο σενάριο το 70% ή πάνω από το χρέος αγοράς που εκρεμεί θα είναι κάτι που είναι πολύ ευάλωτο στην πειθαρχία της αγοράς Πιστεύω λοιπόν ότι ένα παρόμοιο σχέδιο είναι εφικτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική ε, πολιτική για μελλοντικέ καταιγίδε ε, και θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες προς βαθύτερη, μεγαλύτερη εμβάθυνση. Ε, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και γι' αυτό προτείνω αυτό το σχέδιο στην Επιτροπή που σας περιγράφω. Ευχαριστώ πολύ. Ο δεύτερος ανέρα, ο κύριος Βίριελε, Διευθυντής Οικονομικής Έρευνας σε Φινλανδικό Ινστιτούτο. Του δίνω το λόγο για 7 λεπτά επίσης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε μια συγκεκριμένη πτυχή αυτών των ε, εγχειρημάτων που έχει ήδη αναφερθεί από τους προγραλίσαντες αλλά θα είμαι λίγο πιο ε, συγκεκριμένος και θα επικεντρωθώ σε συγκεκριμένους κινδύνους. Ο μερισμός του χρέους μέσω κοινή έκδοσης χρέους έχει βεβαίως ε, επιπτώσει τη συμπεριφορά των ε, αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικής. Και αυτό σημαίνει για τις χώρες οι οποίες θα ωφεληθούν ε, λιγότερη πίεση για, τη βελτίωση, για το στόχο της βελτίωσης της βιωσιμότητας του χρέους. Υπάρχει. Αν θέλετε λίγο πιο γρήγορα. Α, όχι, λίγο πιο αργά. Έχετε την καλοσύνη να μιλάτε πιο αργά, είναι δυνατόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τρόποι να περιορίσουμε τον ε, διοντολογικό αυτόν κίνδυνο. Καταρχάς ε, υπάρχουν και δυνατότητα για χώρες οι οποίες έχουν ε, μόνο πολύ καλό επιδόσεις η δυνατότητα να μπουν στο σύστημα, αλλά βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα περιοριστούν και τα ωφέλη από την αντιμετώπιση, από τον επιμερισμό δηλαδή του κακού χρέους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ αυστηρός έλεγχος της συμπεριφοράς των κρατών μελών από τις ευρωπαϊκές αρχές και δεύτερον τα δημοσιονομικά κίνητρα θα πρέπει να υπάρχουν ενσωματωμένα μέσα στα, στα προγράμματα αυτά κοινή έκδοση. Βέβαια, το ζήτημα το εάν αυτό μπορεί να αρκέσει για να αποτρέψει εσφαλμένη συμπεριφορά. Η οικονομική διακυβέρνηση ήταν αρκετά αυστηρή τα τελευταία χρόνια και είχε αλλάξει σημαντικά την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το six-pack, το πάκ και το Fiscal Compact έχουν συμβάλει σε αυτό. Πριν όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς ο νέος μηχανισμός οικονομική διακυβέρνηση μπορεί να φέρει αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη ε, πολλά περιθώρια να αλλάξει η κατάσταση, δεδομένου ότι πολλά είναι στα χέρια ακόμη των κρατών μελών, άρα θα χρειαστεί αλλαγή τροποποίηση συνθήκης. Ο περιορισμός αυτού του δεοντολογικού κινδύνου μέσω των οικονομικών κινήτρων μπορεί να πάρει διάφορες μορφές ε, με κυρώσεις ως προς τα επιτόκια ή επιβράβευση αντίστοιχα εφόσον υλοποιούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Τελικό στόχο βέβαια πάντα θα είναι η επιδραβευση αντιστοιχα εφοσον υλοποιουνται οι δημοσιονομικοι στοχοι τελικο στοχος βεβαια παντα θα ειναι η πειθαρχια στη δημοσιονομική πειθαρχία και η πειθαρχία στην αγορά αυτό θα πλήττει κράτη-μέλη τα οποία δεν τηρούν τους κανόνες ή δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα για άρνηση πρόσβασης στην κοινή έκδοση, αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να κηρύξει πάυση εξυπηρέτησης των χρεών του, των δεσμεύσεων του ένα κράτος. Το παράδειγμα των Lehman Brothers μας δείχνει ότι, περισσότερο, ότι χρειάζεται περισσότερη ε, πειθαρχία και θα πρέπει να δούμε ότι ο μηχανισμός ESM θα πρέπει να είναι αρκετά στεναρός ώστε να στηρίξει κάθε προσπάθεια προσωρινής ενίσχυσης κρατών μελών. Δεύτερον, θα πρέπει το τραπεζικό σύστημα να είναι σε θέση να αντέξει τη δημοσιονομική αστάθεια που μπορεί να προκύπτει από το κρατικό χρέος. Σε αυτό έχουμε δει σημαντική προόδο κυρίως με τη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά δεν βλέπουμε να έχουν διαραγεί οι δεσμοί μεταξύ κρατικού χρέους και κατάσταση των τραπεζών. Τρίτο και πιο σημαντικό, θα χρειαστεί ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει αναδιάρθρωση, τακτική αναδιάρθρωση του χρέους των κρατών που θεωρούνται αφαιρέγγια. το οποίο δεν προβλέπετε τώρα. Το πρόβλημα με του μηχανισμού είναι ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν από τη μια μέρα στην άλλη, όπω άλλωστε αναφέρθηκε νωρίτερα. Σε μια κατάσταση δηλαδή όπου πολλά κρατημέλη έχουν υψηλό χρέο, τίθεται σε κίνδυνο η στεναρότητα των τραπεζών του. Και άρα φτάνουμε σε μια κατάσταση ότι μπορεί να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες για προφύλαξη σε σχέση με τον κίνδυνο που σχετίζεται με τον επιμερισμό του χρέους. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν ισχυρή πολιτική βούληση για ενίσχυση των μηχανισμών αυτών πριν, μπούμε, πριν αρχίσουν αυτές οι ρυθμίσεις, δεν θα φέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ε, η αντίληψη σε σχέση με τη σοβαρότητα αυτού του δεοντολογικού κινδύνου και των συνεπειών ε, μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Και υπάρχει περίπτωση οι φυστάμενοι μηχανισμοί να ενισχύσουν τον κίνδυνο, κυρίως αν γίνουν οι μηχανισμοί προσαρμογής περιορισμένοι με περιορισμένες εγγύσεις. Ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να θεωρούν τον διοντολογικό κίνδυνο πολύ σοβαρό Αλλά βεβαίω αν προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε ε, αποτελεσματικά την ε, πειθαρχία σε σχέση με τις αγορές, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας Άρα θα πρέπει να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση υπορισμένες προϋποθέσεις επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κρατη και στο σχεδιασμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Επίσης, ε, Υπάρχουν εκείνοι οι υπερογνώμενε που θεωρούν ότι χρειάζεται να περιοριστεί ο διοντολογικό αυτό κίνδυνο και να ενισχυθεί η διακυβέρνηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε ε, όλα τα μέλη του πάνελ των ε, εμπειρογνώμων και τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση με τα μέλη της, ε, Ευρωπα... της Επιτροπής Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να σας πω ότι έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας. Μπορείτε να υποβάλλετε και ερωτήσεις και θα πρέπει να ορίσετε σε ποιον υποβάλλετε την ερώτησή σας, ίσως και σε δύο εμπειρογνώμονες. Αλλά έχετε για πέντε λεπτά το λόγο. Ο κύριος Ζανπόλ ε, Γκοζές από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εγώ θα μιλήσω στα γαλλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες ε, για την ποιότητα της εργασίας τους, γιατί μας δώσαν τα βασικά στοιχεία αυτής της έκθεσης και θα ήθελα να τους συγχαρώ γιατί πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα. Θα έπρεπε να ξεδιαλύνουμε τα τεχνικά ζητήματα από τα πολιτικά για κάθε σύστημα αμοιβεοποίησης του χρέους και νομίζω ότι η εργασία αυτή ήταν πολύ καλή. Φαίνεται λοιπόν ότι μία πραγματική αμοιβεοποίηση του χρέους σημαίνει τροποποίηση των συνθήκων. Αν και άκουσα εναλλακτικές λύσεις που μας επιτρέπουν να λειτουργήσουμε με τις υπάρχουσες συνθήκες. Άκουσα επίσης ότι η θέση σε εφαρμογή μιας τέτοιας αμοιβεοποίησης θα σήμαινε ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης. Και αυτό μας δείχνει ότι τα μέσα αυτής της θητείας του ΠΑΚ, ΣΥΚΣ και Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εφαρμόζονται αυστηρά και συνεπώς οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το κείμενο ε, έχουν αναλυφθεί από τα κράτη. Η ερώτησή μου είναι απλή και περίπλοκη συνάμα. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο κατανόησα σωστά τις ε, συστάσεις της έκθεσης και δεύτερον θα ήθελα να ρωτήσω εάν ε, με βάση τους ε, όρους που προβάλλονται για την αμοιβεοποίηση το θέμα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα επίκαιρο. Ποιος θα απαντήσει. Η πρόεδρος, κυρία Τιμπάλκα. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές για αυτή την ερώτηση. Καταρχήν νομίζω ότι φτάσατε στα, φτάσατε στα σωστά συμπεράσματα. Η κοινή έκδοση είναι ένα μακρόπνο σχέδιο για, τον, για την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ζώνη και μιλάμε για μακρόπνο σχέδια μέσα στα πλαίσια και της αλλαγής των συνθήκων. Πριν κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ κυβερνήσεων και κοινοβουλίων να είναι έτοιμα να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο και τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις και για τα δύο μέσα, για τα επερχόμενα έτη και όχι μόνο με την αρχική σύσταση του σχεδίου κοινής έκδοσης, του κοινού σχεδίου έκδοσης. και κάποιος άλλος από το πάνελ, αν θέλει, μπορεί να απαντήσει, γιατί έχουμε ακόμα δύο λεπτά, αν θέλει. Όχι, ωραία. Περνάμε λοιπόν στον επόμενο, στην επόμενη ομιλήτρια, την Ελίζα Φερέιρα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ το πάνελ των εμπειρογνωμόνων για την άκρος ενδιαφέρουσα και εις βάθος παρουσίαση. Λυπάμαι που δεν είχαμε τα κείμενα νωρίτερα, διότι αυτό θα μας επέτρεπε να δούμε τις λεπτομέρειες και είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιδράσει κανείς άμεσα και σε σχέση με την προεπεξεργασία του κειμένου. Ελπίζω να παραμείνουμε σε επαφή, αν όχι σε αυτή τη θητεία, στην επόμενη. Δηλαδή να προωθήσετε αυτό το διάλογο με το επόμενο κοινοβούλιο στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και αναφέρομαι στην ομιλία της κυρίας Τόπελ Γκούγκερελ Αναφερθήκατε στην κατάσταση πριν δύο χρόνια, πώς συζητήθηκαν τα πράγματα. Αυτή η ομάδα λοιπόν δημιουργήθηκε με αίτημα αυτής της Επιτροπής, δηλαδή από τους ηγητές και σκιώδεις του, Τούπακ και θεωρήσαμε ότι αυτό που συμφωνήσαμε στο μηχανισμό των δύο νομοθετημάτων ήταν κάτι το πολύ δεσμευτικό σε σχέση με τη μακροοικονομική πολιτική μέχρι την, αν όχι την αποπληρωμή, την πληρωμή του 75% του ποσού ε, δανειοληψίας. Αυτά είναι ζητήματα που θέτουν τη διαδικασία σε διαφορετικό πλαίσιο. Μπορούμε να κρατήσουμε τη σταθερότητα της Ευρωζώνης με το υπάρχον επίπεδο χρέους και ρυθμού ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, άλλες εναλλακτικές κάποια λύση για να αντιμετωπίσουμε το διτό αυτό χαρακτήρα, δηλαδή της αιρεσιμότητας του 2-pack και του 6-pack. Δηλαδή πολύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης και χαμηλό επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος. Είδαμε πολλά ζητήματα για τα οποία δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και αναγκαστήκαμε να τα επιλύσουμε. Τώρα αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ε, ε, μπορέσουμε, σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ανταποκριθούμε, ιδιαίτερα στο phasing in. Πώς μπορούμε λοιπόν να ανταποκριθούμε. Ε, όπως είπε ο κύριος Γκρέιμ Μπίσοπ και η κυρία Ανιές και Υπάρχουν άλλα ενδιάμεσα βήματα. Κυρία Αντιμάουρο. υπάρχουν ε, ενδιάμεσες λύσεις για να ε, απομειώσουμε τον κίνδυνο ε, δημιουργίας ή εμφάνισης χρεοκοπίας με βάση την σχετική σταθερότητα στην οποία έχουμε φτάσει τώρα και ποια είναι τα συνιστόμενα βήματα. Το. Από ό,τι κατάλαβα, ε, αποτανθήκατε σε τρεις ή τέσσερις ε, εμπειρογνώμενες, στους οποίους δίνω και το λόγο. Ο, ε, η κυρία Μπενασί και ο κύριος Μπίσοπ. Ο κύριος Μπίσοπ. Με τι ταχύτητα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Σας είπα ότι θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη τον κανονισμό και το άρθρο 352 μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αυτό έχει σημασία, ε, είναι και ε, ο μηχανισμός, η ταχύτητα έγκρισης των ε, νέων συνθήκων, γιατί ο οποιοδήποτε διαχειριστής χρέους θα μπορούσε να το πετύχει αύριο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τις πολιτικές επιπτώσεις και τις νομικές. Και το μόνο πρόβλημα είναι τα εθνικά κοινοβούλια. Αν υπάρχει θέληση μπορούν να εκδοθούν αυτά τα ευρωομόλογα σε ένα χρόνο. Και αυτό αφορά και τις οριστικές νομισματικές συναλλαγές, τα OMTs. Έτσι θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στην έκδοση ευρωμολόγων άμεσα. Η κυρία Μπενασί Κερέ ε, θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ. Θα ε, απαντήσω στο πρώτο ερώτημα Εάν θεωρείτε ότι υπάρχει εξισορρόπηση και ότι η αγορά δεν λανθάνει και ότι δεν υπάρχει ε, πρόβλημα ε, αξιόχρεου, φερεγγιότητας μάλλον, και τα στοιχεία είναι αξιόπιστα, δεν θα αμφισβητηθούν ποτέ από κανέναν, τότε δεν υπάρχει επίγον χαρακτήρας να ορίσουμε νέα μέσα. Ε, αν το σκεφτόμαστε είναι γιατί έχουμε αμφιβολίες για το ένα ή για το άλλο. Ε, αληθεύει ότι τα μέσα που έπρεπε να μας απασχολήσουν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα, γι' αυτό το συζητήσαμε στην ομάδα και συζητήσαμε για πιο ήπιες μεθόδους για να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση χωρίς ε, να ε, βάλουμε ε, τρία τρεις στην παλάντζα. Γι' αυτό μιλάμε για ένα μικρότερο ταμείο απόσβευσης, 20 δηλαδή ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, ε, δηλαδή όχι σε επίπεδο χρέους αλλά σε επίπεδο ΑΕΠ και αυτό ανταποκρίνεται και στις στη κεφαλουχική ανταπόκριση της ΕΚΤ. Θα υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής και θα υπάρχει ρευστότητα η οποία θα μειωθεί. Αλλά η δοκιμή ε, θα δείξει αν πραγματικά αποπληρώνεται το χρέος και έτσι βελτιώνουμε και την αξιοπιστία μας για να μειώσουμε το κόστος αναχρηματοδότησης για τα κράτη χωρίς αλλαγή των συνθήκων, αλλά με ένα καταναλογία σύστημα. Αυτό ακριβώς μας απασχόλησε στην ε, έκθεση. Η κυρία Ντιμάουρο μπορεί επίσης να απαντήσει αν το θέλει. Δέχομαι αυτά που είπε η Ανιές. Ίσως ε, για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, εάν δηλαδή το σχήμα αυτό είναι σχετικό, εν μέρη όχι, διότι ο ε, κατεπήγον μηχανισμός του ΕΚΤ ε, έχει, βγάλει τον, έχει άρει τον κατεπήγοντα χαρακτήρα της καταπολέμησης της χρήσης, αλλά υπάρχει ακόμα η το χρέος, το επικρεμάμενο χρέος και γι' αυτό ίσως οι απαιτήσει του ΤΟΥΠΑΚ να, είναι, να υπάρχουν. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί πρόσκομα για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Άρα ε, υπάρχει ε, επίγον ζήτημα να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτό το Ταμείο Απόσβεσης Χρέους, το οποίο είχε εστιαστεί σε αυτό το ζήτημα. Ε, ο, εκπρόσωπο ο, ο εκπρόσωπος των Φιλελευθέρων, Ράμος Τρεμόζα, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία. Κάποια σχόλια σύντομα για ένα λεπτό και έχω κάποιες ερωτήσεις να υποβάλω. Έχοντας διατρέξει τα συμπεράσματα της εκθέσεως κατά την άποψή μου, τα ευρωμόλογα φαίνονται η πιο ρεαλιστική προσέγγιση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Απόζωσης του Χρέους. Νομίζω ότι ότι δύο προσεγγίσεις μια αναγή συνθήκων θα απαιτηθεί και στο παρόν ε, πολιτικό κλίμα νομίζω ότι χωρίς σαφή λαϊκή εντολή για κάτι τέτοιο στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο δεν βλέπω να υπάρχουν πολλές δυνατότητες να προχωρήσουμε σε αυτά. Άρα, αν υπάρχει πολιτική βούληση για κάποια κράτη-μέλη, αυτά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να περάσουν μέσω διεργασίας, διευρυμένης συνεργασίας και διακυβερνητικής συμφωνίας. Νομίζω ότι αυτό το τελογικό κίνδυνος πρέπει να αποφευθεί και ρεσιμότητα απαιτείται. Το ερώτημα είναι τι είδους ρεσιμότητα θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, οι χώρες θα πρέπει να, να ισολογίζουν τον προπολογισμό τους ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρεμβαίνει στον προπολογισμό των κρατών μελών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Πόσο πρέπει να ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον προπολογισμό των κρατών μελών για να αποφευχθεί αυτό ο δεντρολογικός κίνδυνος. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και τέλος, ε, έχετε κάποιες πληροφορίες, τι αντίδραση έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αφορά τις προτάσεις σας. Τελευταίες δύο ερωτήσεις. Αν τα ευρωομόλογα είχαν εφαρμοστεί πριν από την κρίση, ποια θα ήταν αντίκτυπος στα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά. Μπορείτε να εκτιμήσετε λίγο πολύ αυτό τον αντίκτυπο. Για κάθε χώρα που πρέπει να ε, αντιμετωπίζει κρίση, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ποιος απαντά σε αυτές τις άκρως ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση όσον αφορά το είδος της αιρεσιμότητας. Απαιτείται όσο πιο πολλές χώρες δέσουν τις μοίρες τους με τις άλλες, θέλουν να έχουν διαβεβαιώσεις και ελέγχους ότι μπορούν να παρέμβουν αν τα πράγματα πάνε στραβά. Γι' αυτό Μία από τις δυνατότητες είναι να μην παραμένει εθνική κυριαρχία σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αυτό που συζητήσαμε ήταν συμπροματική εξουσία παρέμβαση στις εθνικές πολιτικές να χορηγείται αν δεν τηρούνται υποσχέσεις επανειλημμένα δεν είναι μόνο αν υπάρχει απόκληση μία φορά, αλλά αν δεν υπάρχει συμμόρφωση επί μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε κάποιε απαντήσει, κάποιε αντιδράσει. Θα ήταν ε, ενδιαφέρον να έχουμε κάτι τέτοιο. Συνεργαστήκαμε στενά με εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας έδωσαν ε, υποστήριξη πλευρά γραμματείας, αλλά δεν έχουμε κάποια αντίδραση όσον αφορά Όσον αφορά τις οικονομίες, έγιναν πολλές συζητήσεις κατά πόσο θα μπορούσαμε να κάνουμε υπολογισμούς για ενδεχόμενες οικονομίες. Στο τέλος όμως προτιμήσαμε να περιγράψουμε τάσεις, ενδεχόμενες ε, επιπτώσεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε μελλοντική τιμολόγηση του κρατικού χρέους, διότι αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν θα ήταν σοβαρό να δώσουμε ποσοτικοποιημένη απάντηση όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνέπειες, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μπίσοπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ να σχολιάσω την ερώτηση για τα ευρωμόλογα. Αν αλλαγή των συνθήκων είναι κάτι που απαιτείται. Στην πρότασή μου δεν απαιτείται. Με την πάροδο του χρόνου, αν όλα πάνε καλά και ανοίξει για άλλους σκοπούς αυτό το ταμείο, ε, θα μπορεί να βασιστεί στο, στη συνθήκη το Ταμείο. Για την ώρα, μια κυβερνητική απόφαση για τη λήψη αποφάσεων μεταξύ κρατών μελών για το πόσο δανείζεται ο κόσμος, που είναι κάτι εκτός της συνθήκης, και όλα τα άλλα. Η διαχείριση του χρέους, η υπηρεσία διαχείριση του χρέους, όλα αυτά μπορούν να γίνουν δυνάμει του άρθρου 352, μέσω κανονισμού της κοινότητας. Δεν απαιτείται μια τροποποίηση των συνθήκων. Euh, Πάμε τώρα στον επόμενο μιλητή, ECR, ο κύριος Τρέσεκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, πόσο χαριτωμένη αλλαγή στην Προεδρία, κυρία Πρόεδρε. Και είσαστε τόσο ευγενικοί ίσως μου δίνετε και περισσότερο χρόνο να, αν είμαι ευγενικό να θέσω ερωτήσει. αλλά όχι, όχι. Ευχαριστώ πολύ για την λεπτομερή παρουσίαση από πλευράς όλων των εμπειρογνωμόνων. Βλέποντας τις παρατηρήσεις μου, βλέπω τρεις βασικές παρατηρήσεις που έχω σημειώσει. Τρία σημεία, τα οποία ανέφεραν κατά κάποιο τρόπο ο καθένας από εσά, οδολογικός κίνδυνος, νομικές απαιτήσει και ενδεχόμενες ε, τροποποίησεις, αλλαγές των συνθήκων. Όντας ανοιχτός, ειλικρινής και δίκαιος, θα έλεγα ότι η θέση του ECR κατά τη διάρκεια των συζητήσεων περιστρέφεται γύρω και από τα τρία σημεία τα οποία θίξατε και εγώ θέλω να σας ζητήσω να ξεκαθαρίσετε περισσότερο τις θέσεις σας. Αυτή θα ήταν η, τάση μου, αλλά καταλαβαίνω ότι οι απαντήσεις όσον αφορά τα σχόλια αυτά βασίζονται στην προθυμία των κρατών μελών να παρετηθούν από ορμοδιότητές τους υπέρ της προτάσεως που συζητούμε και περιγράφεται. Η ερώτησή μου λοιπόν δεν θα βασίζεται επί του δοντολογικού κινδύνου και των νομικών απαιτήσεων και των αλλαγών των συνθήκων και είναι η εξής. Όσον αφορά τα προτινόμενα ευρωομόλογα τα οποία μπορούν να περιγραφούν σαν ομόλογα με βραχυπρόθεσμη ορίμανση, οριμότητα. Μπορούν να ξεκαθαρίσουν οι απαΐοντες, ίσως η κυρία Πρόεδρος των ε, ποια είναι η, ενδεχό, η απόδοση, η αναμενόμενη απόδοση των ευρωομόλογων και τι είδου εγγύηση απαιτείται, για την αξιοπιστία τους και την πιστοτική τους, πιστοληπτική τους ικανότητα στις αγορές. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Τολμάτε να δώσετε τις απαντήσεις πρώτοι, όπως σας ζήτησε ο κύριος Βουλευτής, η κυρία Πρόεδρος. Έχετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για, την... για τους πιθανούς υπολογισμούς του κόστου της χρήσης. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν διαφέρει πολύ σε επιτόκιο ε, το ευρωπαϊκό ομόλογο, άρα είναι πολύ κοντά τα επιτόκια και έτσι ως συνέπεια θα περιμέναμε όχι τόσο τιμολογιακή αλλά περισσότερη διάδοση των ομολόγων, μεγαλύτερη αγορά δηλαδή των, αγορο των ομολόγων και άρα πιο σταθερή αγορά. Και το δεύτερο, αν θέλετε να μου επαναλάβετε το δεύτερο τμήμα της ερώτησης, οι εγγύησεις. Εμεί βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα χρειαστεί κεφάλαιο ως βάση της ε, πολιτικής του και θα αρκούσε αυτό το κεφάλαιο. Έχουμε συστήσει επίση το θέμα πιθανών εγγύσεων, χορήγηση πιθανών εγγύσεων, αλλά φαίνεται να είναι αρκετά περίπλοκο αυτό να εξασφαλιστεί, δηλαδή να σύστημα εγγύσεων για τι διάφορε χώρε. Δεν είναι δυνατόν εύκολα δηλαδή να ποσοστοποιήσουμε. Και άρα μάλλον η χορήγηση κεφαλαίου με βάση το ESM δεν είναι η καλύτερη λύση. Αν μου επιτρέπετε να κάνω κι εγώ μια παρατήρηση για την αναμενόμενη απόδοση τουλάχιστον τα δύο τρίτα αυτών των ομολόγων θα τα διακρατούν τράπεζες, θα επαναχρηματοδοτούν δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυτό θα είναι κυρίως, αυτός θα είναι κυρίως ο μηχανισμός επανατροφοδότησης. Αυτή πιστεύω ότι θα είναι η κύρια επίδραση. Και μια και θα έχουμε έλτρο διετή, πιστεύω ότι αυτό θα είναι η, η κινητήρια δύναμη. Ευχαριστώ πολύ και περνώ στον επόμενο μιλητή. Ο κύριος Λάμπερτς εκ μέρους της ε, ομάδας των Πρασίνων. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω τρει σύντομε ερωτήσει προ του ε, ειδικού εδώ, ποιος θέλει να απαντήσει. Νομική και τεχνική η πρώτη ερώτηση, νομοτεχνική ούτω η είναι. Μα λέτε ότι χρειάζεται κανονισμό του 352 και διακυβερνητική συμφωνία. Ο κύριος Μπίσοπ νομίζω έδωσε την απάντηση, αλλά θα ήθελα να μου εξηγήσει περισσότερο γιατί χρειάζεται διακυβερνητική συμφωνία για το μηχανισμό αυτό. Ε, και βέβαια αυτό συγκρινόμενο με την απόφαση, σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για δε ρύθμιση του τύπου Euro Rates, δηλαδή επανασταθεροποίηση των επιτοκίων και αναδιανομή του ωφέλους εκείνων που δανείζονται με χαμηλό επιτόκιο προς εκείνους που έχουν επιβαρυνθεί με πιο υψηλά επιτόκια. Επίσης, μια και ζω σε πραγματική χώρα, και βλέπω ότι τα μεγάλα δεν ε, σέβονται τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης, ούτε αυτά. Και επίσης μια και κάποιος από εσά ανέφερε ήδη ότι ε, ο λόγος χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ αυξάνεται σχεδόν παντού. Δεν θέλω να μου πείτε εσείς, ποιο ήταν το κόστος της μη εφαρμογής από αυτά τα μέτρα. Γιατί ακούω από αυτά που μου λέτε ότι υπενήσεστε πως καλό θα ήταν να γίνει το ένα και το άλλο, αλλά θα μπορούσε και να μην γίνει τίποτα και δεν πειράζει. Και εδώ ήταν το κόστος λοιπόν για την Ευρώπη. Εάν δεν υλοποιούνταν τίποτε στον χώρο της αμοιβοποίησης του χρέους, είτε πρόκειται για το παρελθόν είτε πρόκειται για το μέλλον χρέους, θα ήθελα να ρωτήσω εάν πράγματι ε, θεωρείτε ότι μπορεί να κινδυνεύει το ευρώ, Φερρυπίν. Ευχαριστώ πολύ. Μας μένουν μόνο τρία λεπτά. Σας παρακαλώ να είστε σύντομη η Πρόεδρος. Για την πρώτη ερώτηση θα απαντήσω εγώ, ίσως ένας άλλος συναδέλφος να θέλει να απαντήσει τη δεύτερη. Γιατί χρειάζεται ο συνδυασμός κανονισμού και διακυβερνητική. Δεν θα είναι αρκετή η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό δίκαιο αν δεν γίνει τροποποίηση συνθήκης. Αυτό βασικά. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό προτείνουμε κανονισμό μαζί με διακυβερνητική συμφωνία. Για το δεύτερο ερώτημα, ποιος θέλει. Κοιτάξτε, δεν συζητήσαμε ιδιαίτερως την πρόταση αυτού του euro για τα, για τα επιτόκια δηλαδή, εξίσωση των, των επιτοκίων. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν, μπορούμε να αναμένουμε ότι θα παρακολουθήσουν τη ρύθμιση της κατάστασης και άρα μπορούν να έχουμε αντίστοιχα ε, προβλήματα στην υλοποίηση όπως αυτά της κοινή έκδοσης. Για τελευταία σας ερώτηση δε, ποιο είναι το κόστος εάν δεν επιμεριστεί καθόλου το χρέος. Ε, αυτό που θα απαντήσω είναι ότι δεν έχει να κάνει ή δεν μπορεί αποτελεσματικά να καταπολεμήσει το εκρεμές χρέος αυτή η πρόταση γιατί το κόστος της χαμηλής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι πολύ υψηλό. Τώρα, εάν η, ο επιμερισμός του χρέους είναι η μόνη λύση, μάλλον όχι, αλλά ίσως, να, μην είναι, ίσως να και χειρότερος, να είναι καλύτερη. Από την άλλη, κύρια προτεραιότητα είναι να περιοριστεί το ε, εκρεμές και ληξιπρόθεσμο χρέους και αυτό πρώτα απ' όλα πρέπει να εξεταστεί. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Non, évidemment que ça ne va pas. Je veux dire, tout ça est bien gentil, mais enfin... Όχι, όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Ε, ε, πολύ ευγενική, πολύ σπαθή μου είστε και όλα αυτά, αλλά αν μου λέγατε κάτι τέτοιο σε ένα διαγώνισμα θα σα έκοβα ω καθηγητή. Το να μου λέτε ότι κάνουμε τη διακυβερνητική γιατί καλό θα είναι να υπάρχει διακυβερνητική. Δηλαδή και εγώ θα μπορούσα να απαντήσω, να συνεχίσω με την ε, λεγόμενη ταυτολογία. Ε, μου λέτε ότι πρέπει να κάνουμε διακυβερνητική γιατί πρέπει να γίνει διακυβερνητική. Ε, Πείτε μου, από τις συνθήκες τι είναι αυτό που εμποδίζει ε, την έκδοση ενός κανονισμού που να ρυθμίζει. Αλλά μέχρι τώρα έχετε κοπεί, είστε κάτω από τη βάση. Η Πρόεδρος. Ναι, και εγώ θέλω να ακούσω την απάντηση. Ο κύριος Μπίσοπ νομίζω ότι είχε μια λύση να προτείνει χωρίς τροποποίηση των συνθήκων. Η Πρόεδρος πρώτα. Χωρίς μικρόφωνο όμως. Οι νομικοί δικηγόροι με τους οποίου μιλήσαμε μας είπαν ότι οι αρμοδιότητε όπω αυτέ καταγράφονται στη συνθήκη αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν για να θεσπιστεί ένα τέτοιο σύστημα. Εάν θέλουμε λοιπόν τέτοιο σύστημα θα πρέπει να γίνει να εξασφαλιστούν πρόσθετα νομοθετήματα. Και άρα η ιδέα της, ε, του συνδυασμού μιας κυβερνητικής συμφωνίας μαζί με τα σχετικά άρθρα της συνθήκης θεωρήθηκε ένας τρόμος, μια λύση, χωρίς αυτό να, σημαίνει ότι πρέπει να πάμε αμέσω σε αλλαγή συνθήκης, για να μην πάμε σε αλλαγή συνθήκης αμέσως. Κύριος Μπίσοπ, ναι, κοιτάξτε, το κέριο στοιχείο εδώ είναι ότι η συνθήκη όπως ισχύει μιλάει για συντονισμό οικονομικής και δημοσιονομική πολιτική. Ενώ εγώ μιλάω για μια πρόταση από τα κράτη-μέλη, από τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη, ώστε να μην εκδίδουν βραχυπρόθεσμα ομόλογα, αλλά του ευρωομολόγου. Αυτό νομίζω ότι είναι η λύση. Και σε αυτό ήταν σαφές ε, ε, από τους ε, δικηγόρους, τους πραγματογνώμονες νομικούς, ότι δεν γίνεται να μην τροποποιηθεί η συνθήκη εφόσον επιδοκόμενος στόχος είναι αυτός. Γι' αυτό μιλούμε για διακυβερνητική. Κύριος Λάμπερτς, το τελευταίο ήταν κάπως πιο συγκεκριμένο. Περνάτε, η συνάδελφός σας όμως παραμένει κάτω από τη βάση. Γιατί όταν μου λέτε μου είπανε ότι δεν μου αρκεί η απάντηση. Ο κύριος Κλουτα. Πολλά συγκεκριμένα ερωτήματα έχουν διατυπωθεί. Εγώ θα ήθελα να περάσω σε ένα πιο πολιτικό επίπεδο. Από την αρχή του έτους μια αντιπροσωπεία μας επισκέφθη τα κράτη που αντιμετωπίζουν κρίση και εγώ έχω την εντύπωση, από αποκομίσει, ότι η κρίση όπως εξελίσσεται έχει πολύ μεγάλο, ενέχει πολύ μεγάλο πολιτικό κίνδυνο. Ιδιαίτερα για την Πορτογαλία, βλέπω ότι είναι η κατάσταση πάρα πολύ κρίσιμη, το ίδιο και για την Ελλάδα, πολιτικά κρίσιμη. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ εάν μπορούν να βρεθούν άλλες εναλλακτικέ. Και δεν βλέπω με δεδομένο ε, αυτό το κατεπήγον της ανάγκης γιατί δεν αναζητούμε και άλλες εναλλακτικέ. Και μια ερώτηση για σας. Εάν τα προτινόμενα μέσα αυτά που συζητούμε τώρα δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν αμέσω, τι εναλλακτική θα είχατε να προτείνετε. Κάτι ακόμη, πολύ σύντομα. Έγινε λόγος για κίνητρα που οδηγούν στο αντίξω αποτέλεσμα. Ναι, βεβαίως, συμφωνώ και εγώ ότι δεν πρέπει να ε, προξενήσουμε περισσότερη κρίση με τα κίνητρα αυτά. Από την άλλη όμως, ε, το υπερβολικό χρέος στα κράτη δεν μπορεί απλά και μόνο να αποδοθεί σε υπερβολικές κρατικές δαπάνες. Η κρίση του ε, τραπεζικού τομέα, του χρηματοπιστωτικού εν γέννη τομέα ήταν αυτή η οποία οδήγησε στη μεγάλη κρίση. Μπορώ να δεχθώ ότι στην Ελλάδα, και αυτό είναι αναμφίβολο πιστεύω, υπήρξαν και άλλοι εσωτερικοί λόγοι που επιδίνωσαν την κρίση, αλλά η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη, δεν μπορούμε να την, ε, να την ε, αναγάγουμε, να την υπαγάγουμε μάλλον σε κάτι τόσο απλό. Άλλωστε δεν ξέρουμε και το ρόλο της Γερμανίας σε όλο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε τι είδους αναλλακτικέ βλέπετε εσείς. Ίσως ε, και άλλα μέλη της Επιτροπής μπορούν να απαντήσουν. Η δύσκολη πολιτική λύση ανακύπτει γιατί ε, εφαρμόστηκαν μακρόπνοες πολιτικές, αλλά ε, υπήρχαν, ε, μάλλον προβλήθηκαν πολιτικές λύσεις πολύ συσταλτικές, πολύ περιοριστικές. Αυτό σε σχέση με τις δημοσιονομικές πολιτικές που προβλήθηκαν μερικά χρόνια πριν μπορεί, δηλαδή να καταπραϊνθεί η κατάσταση, αλλά όχι ολιστικά. Ως προς τις ε, Εναλλακτικέ. θα ήθελα να πω ότι τα παραδοσιακά σχέδια δεν είναι μία μαγική λύση. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μία πολιτική ε, συνένεση για το κατά πόσο πραγματικά επιθυμούμε μία μεγαλύτερη ολοκλήρωση, ναι ή όχι. Έχετε τώρα. Θα απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις για το κόστος της μη εφαρμογής για την παρούσα κατάσταση, η οποία είναι απαράδεκτη. Θα πρέπει να ε, ποσοστοποιήσουμε την ε, κρίση, να δούμε ποιο είναι το κόστος ε, της κρίσης, πώς μπορούμε να βγούμε από αυτήν και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία νέα διαχείριση με βάση τα μέσα που έχουμε. Με βάση δηλαδή το, τη σταθερότητα και το OMT. Μετά το θέμα είναι καθαρά ε, προσωπικής κρίσης. Το κόστος είναι πολύ υψηλό. Εάν αντιμετωπίσουμε μία νέα κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, χρειάζεται να γίνει ε, bailout, χρειάζεται διάσωση. Αλλά το κόστος αυτό μειώνεται ε, με βάση τα μέσα που προβάλλουμε. Πιστεύω δηλαδή Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μπορούμε να κρίνουμε τη συμπεριφορά των κρατών και τη δυναμική τους, γιατί βρίσκονται σε ένα μεγάλο νεφέλωμα. Η έκθεση θα πρέπει να είναι πηγή ιδεών για ε, την περίπτωση που θα ανακύψει εκ νέου αυτός ο κίνδυνος σε κάποιο κρατός μέλος. Θα πρέπει να προσέχουμε όταν ε, ποσοστοποιούμε μία ε, τέτοια σχέση στην περίπτωση που υπάρχει αποπληρωμή χρέους. Ε, είναι όμως πολύ ρόδινο αυτό το σενάριο για να το χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς, ως benchmark. Ε, δυστυχώς ε, τα σενάρια είναι πολύ πιο ζωφερά και οι λύσεις φυσικά ενέχουν ένα συγκεκριμένο κόστος. Θα πρέπει όμως να συγκριθεί με άλλες λύσεις που είναι επίσης δαπανηρές. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω τώρα ότι ε, ε, έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Η κυρία Τάισεν, ο κύριος Αντολίν Σάντσες Πρεζέδο για τους σοσιαλιστές, η κυρία ε, Ποδηματά, η κυρία Περβάνς και ο κύριος Όλε Σμιτ από τους φιλελεύθερους. Υπάρχουν άλλα ε, μέλη που θέλουν να παρέμβουν, είτε από το ΕΛΚ, ο κύριος Γκίγκολντ. Και εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος του ΕΛΚ. Λοιπόν, πέντε λεπτά έχετε ο καθένας. Η Μαριάν Τάισεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες και τους εισηγητές για τις πληροφορίες που μας έδωσαν, αλλά αυτό που αποκομίζω είναι ότι δεν φτάσαμε σε καμία συμφωνία. Ε, ο κίνδυνος δεοντολογίας υφίσταται, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη πειθαρχία. Αυτό απαιτείται από τα κράτη-μέλη Περιμένουμε αυτή την πειθαρχία εδώ και καιρό και θα πρέπει να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για αυτή την πειθαρχία, όπως έγινε και με τα six pack και 2 pack. Ε, ακολουθούμε τις ίδιες ε, γραμμές, αλλά χρειάζεται να διαθέσουμε πολλά χρήματα και δεν μπορούμε να δεχτούμε την απώλεια νομικής ασφάλειας θα πρέπει να υπάρχει μία εγγύηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν υπάρχει. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες, όποιος ε, νομίζει ότι του αποτείνεται η ερώτηση μπορεί να απαντήσει. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε πίσω την κατάσταση, πίσω μας δηλαδή να έχουμε μια πιο ήπια αντιμετώπιση, μια ήπια αμοιβεοποίηση έτσι ώστε να δούμε τι θα επιτύχουμε βράχη και μέσο πρόθεσμα. Γιατί θα πρέπει να βρούμε τις ρίζες της κακοδαιμονίας, να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ένα ταμείο απόσβεσης του χρέους και να ε, δούμε κατά πόσο ένα τέτοιο σχήμα είναι βιώσιμο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην οδό της αμοιβεοποίησης, αλλά αυτό θέλουμε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να βρούμε μία μακροχρόνια λύση. Τι θεωρούν ότι πρέπει να κάνουμε οι εμπειρογνώμονες. Θεωρούν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα πειθαρχία που έχουμε στη διάθεσή μας και να δούμε κατά πόσο θα έχουμε ένα καλύτερο ταμείο, το οποίο θα έχει συσταθεί σωστά. Εάν οι εμπειρογνώμονες ε, με βάση την ε, έρευνά τους και τις γνώσεις τους ε, κρίνουν ότι υπάρχει κάποια άλλη, κάποιο άλλο μέσον που δεν αντιμετωπίσαμε μέχρι τούδε, ίσως θα ήταν ένας τρίτος δρόμος. Έχουμε εναλλακτικές ε, ενός ε, ταμείου απόσβεσης χρέους ή τίποτα. Αυτό είναι το δίλημα που αντιμετωπίζουμε. Regarding the first question... Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, θυμόσαστε πόσα χρόνια χρειάστηκαν για την θέσπιση της ΟΝΕ και πολλές πτυχές της δεν είχαν προβλεφθεί. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να προετοιμάσουμε μια τέτοια κίνηση. Επίσης ε, συζητήσαμε και το θέμα των δυνατοτήτων, το δυνατοτήτων μας σε σχέση με ιδιωτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς. Η αγορά δημιουργεί διάφορα ε, μέσα αντιμετώπισης ανάλογα με τη χώρα αλλά δεν το συζητήσαμε εις βάθος. Ίσως θα ήθελαν και άλλοι συνάδελφοι να σχολιάσουν. Ο κύριος Βιρέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα κατά πόσο πρέπει να κινηθούμε τώρα, να λάβουμε δράση τώρα ή να περιμένουμε και να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο παρόν μηχανισμός διακυβέρνησης. Είναι δίκοπο μαχαίρι στον κίνδυνο. Αν δεν δράσουμε τώρα, το πρόβλημα του επικρεμάμενου χρέους ίσως να αυξηθεί σαν πρόβλημα για την, και να δημιουργεί κινδύνους για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, κυρίως αν έχουμε και άλλους κλειδονισμούς στο μέλλον. Το να διατηρήσουμε το πρωτογενές πλεόνασμα ίσως είναι πολύ δύσκολο για κάποιες χώρες. Υπάρχουν κίνδυνοι. Απ' την άλλη τώρα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλα τα μέτρα που θέλουμε να θεσπίσουμε κατά του διδολογικού κινδύνου θα πρέπει να υπάρχουν όταν θα εισάγουμε οποιαδήποτε αμοιβεοποίηση. Διότι προσπαθώντα να το θεσπίσουμε αυτό εκ των υστέρων και να διορθώσουμε τα πράγματα είναι δυσχερέστατο. Εν αυτή τη ενία λέγω, αν θέλουμε να προχωρήσουμε αμέσω, θα πρέπει όλο το πακέτο να προωθηθεί. Όλο μαζί. Thank you. Um, I, I can foresee a Προβλέπω μια αλληλουχία γεγονότων. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με προσωρινό ταμείο με βρομόλογα που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και γρήγορα. Και μετά από κάποια περίοδο, όταν αποφασίσουμε να αλλάξουμε τη συνθήκη, μπορούμε να σκεφτούμε και το Ταμείο Απόσβαση του Χρέου. Και το τρίτο στοιχείο που σίγουρα θα πρέπει να το εξετάσουμε και το σκεφτούμε είναι το θέμα τη πειθαρχία τη αγορά που θα εφαρμόζεται στι τράπεζε και στι ασφαλιστικέ ζωή που έχουν στα χέρια του κρατικό χρέο. Κάτι που είδαμε σαφώς όταν έκανα την έρευνα είναι και το εξής. Ο βαθμός στον οποίο εσείς αυτή την Επιτροπή θέσατε όρια εκθέσεως 25% του κεφαλαίου στις τράπεζες που δανείζουν οποιοδήποτε δανειζόμενο εξαρτάται από τα κράτη-μέλη έχουν 50% του κεφαλαίου τους που έχουν δανείσει κάτω από δύο χρόνια και άλλο 100% που το έχουν δανείσει για παραπάνω από δύο χρόνια. Με άλλα λόγια, 150% του κεφαλαίου τους έχει δανειστεί στην κυβέρνησή τους τα κράτη-μέλη. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος που πρέπει να σταματήσει. Και αυτό θα πρέπει σταδιακά να γίνει, θα πρέπει να, να βρεθεί σε μια τρίτη, τρίτος δρόμος του μηδενικού κινδύνου. Είναι μια τρίτη πτυχή που υποχρεώνει τις κυβερνήσεις σε πειθαρχία τη αγορά. Το 70% του κρατικού χρέου που δεν είναι σε προσωρινό ταμείο των ευρωμολόγων θα εκτεθεί στην πειθαρχία της αγοράς. Εάν δεν μπορείς να γεμίσεις τις τραπεζέ σου με αυτό θα πρέπει να το μοιράσει το χρέο στους αποταμιευτές της Ευρώπης και αυτό θα είναι συνεχές δημοψήφισμα θα έλεγα. Είναι πολύ ισχυρή δοκιμή αυτή, πολύ δύσκολη δοκιμή. Ε, I wanted to mainly um, answer... Θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις για εναλλακτικέ και αν σκεφτήκαμε εναλλακτικέ εντός της εντολής της εκθέσεως εξετάσαμε ακροθυγώς απλώς εναλλακτικέ. Αλλά είναι προφανές ερώτημα και σημαντικό και θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν εναλλακτικέ βέβαια για τη μείωση του επικρεμάμενου χρέους μέσω της αμοιβαιοποίησης είναι το μονοπάτι της αμοιβαιοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο μονοπάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει τα επιτόκια και το κόστος χρηματοδότησης είναι μια επιχείρηση εγχείρημα ροής. Υπάρχουν προτάσεις που θα επιτρέψουν ε, λύσεις χωρίς αμοιβαιοποίηση και θα πρέπει να προσημειωθεί όμως εισόδημα φορολογικό και θα καλυφθεί το χρέος ταχύτερα συντονισμένα σε κάθε χώρα είναι η πρόταση πάντρε όπως αποκαλείται και μεταβλητές που δεν εμπλέκουν απαραίτητα την ΕΚΤ. Όσον αφορά το να υπάρχει ασφαλέ στοιχείο ενεργητικού, υπήρχαν κάποιε άλλε προτάσει που, που μέσω, και απαιτούν αμοιβεοποίηση μέσω διάθρωση και ομαδοποίηση εθνικών χρεών κρατών χωρί κοινή έκδοση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε ότι υπάρχουν εναλλακτικέ. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν διαθέτουμε εναλλακτικέ. Υπάρχουν εναλλακτικέ. Ιδού συμπληρωματική όσον αφορά τις εναλλακτικέ. Εντός της ομάδας συζητήσαμε και πρόταση που έκανα εγώ για συμπληρώμαση του μηχανισμού σταθεροποίησης να γίνουν πιστοτικέ τα κονδύλια υποχρεωτικά από τη στιγμή που συμμορφώνεται μια χώρα με τη διακυβέρνηση, έχει αυτόματη πρόσβαση σε πίστοση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίηση και αυτό εξομαλύνει την πρόσβαση στο Μηχανισμό Σταθεροποίηση σε περίπτωση κρίση. Μετά από μια περίοδο το πρόγραμμα σταθεροποίηση γίνεται υποχρεωτικό. Άρα έχουμε ένα εργαλείο σταθεροποίηση χειρίσεω του κινδύνου. Είναι ευρωομόλογα ανάγκη, όπω τα αποκαλώ. Γέφυρα μεταξύ τη κανονική καταστάσεω και πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίηση. Για να μην για να σταματήσουμε αυτή την ασυνέχεια μεταξύ του, ε, της ομαλής καταστάσεως και της προσφυγής των Ευρωπαϊκών Μηχανισμών Σταθεροποίησης. Ο κύριος Σάντσες Πεσέιντο είναι επόμενο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να είχαμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις πριν από την τελική έκθεση, γιατί το θέμα αυτό ε, ήταν πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Θα ήταν ε, σκόπιμο λοιπόν να είχαμε τα δεδομένα αυτά πριν. Το θέμα της, του δεοντολογικού κινδύνου είναι ε, ένα υφιστάμενο θέμα, υφιστάμενο θέμα, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, από ε, μακροοικονομικής πλευράς πώς θα αντιμετωπίσουμε το χρέος, γιατί υπάρχει το κρατικό χρέος, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπτώσεις στο δημόσιο κορβανά. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και μία καθαρά νομισματική πολιτική, ίσως μονεταριστική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό. Μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επίπεδο του χρέους και να δούμε ε, παρά τον όγκο της, ε, κατά πόσο μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Εδώ ε, μιλάμε για έναν δεοντολογικό επίσης κίνδυνο που είναι και αναδρομικός, δηλαδή είδαμε πού ακριβώς αποτύχαμε. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί απάντηση σε αυτό το σκέλος του προβλήματος και να ρωτήσω μέσα στα πλαίσια του Δημοσιονομικού Συμφώνου, του Fiscal Compact, ποια είναι τα μέσα που πρέπει να προωθήσουμε για την μακροοικονομική διακυβέρνηση. Έγινε λόγος για διάφορες εναλλακτικές, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Χρειάζονται όμως άμεσες λύσεις, διότι λειτουργούμε με ε, μεγάλη βραδιπορία και θα πρέπει να βρούμε λύσεις ε, και πιο μακροχρόνια. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής ε, δημοσιονομικής προσέγγισης του όλου θέματος για να αντιμετωπιστεί και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σε ποιον να δώσω το λόγο. Στην Πρόεδρο. Λοιπόν, το πρώτο σημείο. Όσον αφορά το θέμα αυτό, θέλω να πω το χρονοδιάγραμμα ήταν στην ερώτηση. Τι χρονοδιάγραμμα θέλουμε. Α, γυρίσω στα αγγλικά, λέει η πρόεδρος. Και συνεχίζει τα γερμανικά. Πράγματι, σε περίπτωση κρίσης δεν έχουμε, τη στιγμή της κρίσης δεν είχαμε την πλήρη ολοκλήρωση της χρηματοδοτικής αγοράς και δεν προχωρήσαμε αρκετά. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι το σύστημα και τα εθνικά οικονομικά τελικά αποσυνδέθηκαν το ένα από το άλλο και αυτό οδήγησε σε μια ε, αύξηση της κρίσεως. Πρέπει να φτάσουμε στην περίπτωση, στην κατάσταση κατά την οποία έχουμε καλύτερη διασύνδεση αυτών και στην περίπτωση των κρατικών χρεών να μπορούμε να έχουμε ένα σταθερότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να πιέζονται λιγότερο οι κυβερνήσεις έτσι. Νομίζω ότι θα πρέπει το θέμα της ολοκληρώσεως να το βάλετε στη μέση του προβληματισμού σας, στο επίκεντρο. Και θα πρέπει το χρηματοπιστωτικό σύστημα να εξετάζεται σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Το όλο ζήτημα της αλληλουχίας είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε. Πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις. Η, ε, η αμοιβιοποίηση της διαδικασίας θα βοηθούσε. Θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας επίσης ότι η αμοιβεοποίηση του κινδύνου σημαίνει ότι τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παίξουν ε, σημαντικό ρόλο στο μοίρασμα του, του κινδύνου, στην αμοιβεοποίηση του κινδύνου και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι προσεγγίζουμε το θέμα αυτό με το σωστό χρονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Μπέναση, να συμπληρώσω κάτι. Στην ομάδα συζητήσαμε μόνο το, το θέμα των χρεών που κληρονομούνται, Και μετά έχουμε και το θέμα του φορολογικού δυναμικού που βλέπει προς το μέλλον περισσότερο, δηλαδή να υπάρχει ε, για νέα προγράμματα αποταμίευση ε, για, σε επίπεδο ευρωζώνης. Δεν το συζητήσαμε αυτό. Αυτό που απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πολιτικό περιθώριο για τις ιδέες αυτές ή αν υπάρχει συμπληρωματικότητα ή αντικατάσταση. Το ένα σχέδιο αντικαθιστά το άλλο. Δεν έχω απάντηση. Σίγουρα μιλάμε για μεγάλα ποσά Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν συζητούμε τα στοιχεία ενεργητικού να μην καλύπτουμε όλο το περιθώριο της συνεργασίας αν θέλουμε παράλληλα να εισαγάγουμε και ένα δυναμικό φορολογικό που αν θέλετε θα βασίζεται και σε ένα επίπεδο αλληλεγγύης. Um, Ίσως ένα σχόλιο για αυτό το δυναμικό που, που σχετίζεται και με το τι γίνεται μακροπρόθεσμα και ποια είναι η ιδέα της σταθερής πλεύσης αν θέλετε, steady state και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που κληρονομούν το παρελθόν και πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί στο μέλλον ο μηχανισμός σταθεροποίησης. Τι εφαρμόζεται σε κεντρικό, τι σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το δυναμικό, το οικονομικό είναι μια δυνατότητα μοιράσματος του κινδύνου μακροπρόθεσμα αλλά συμπληρωματικό στοιχείο θα μπορούσε να είναι ένα καθεστώς αναδιάθρωσης που εξελίσσεται εφαρμόζοντας δημοσιονομική πειθαρχία σε εθνικό επίπεδο και μπορεί να είναι ένα άκρο σταθεροπιστικό στοιχείο στα δεύτερη γραμμή άμυνας πίσω από όλα τα μέτρα διακυβέρνησης που έχουν θεσπιστεί εάν σχεδιαστεί σωστά βέβαια. Βέβαια δεν μπορεί να σχεδιαστεί ούτως ώστε να δημιουργεί άμεσα διαταράξεις, θα πρέπει να σχεδιαστεί με έναν τρόπο που οι χώρες να είναι κάτω από το όριο και να ενθαρρύνονται να μένουν κάτω από το όριο και να λαμβάνει η χώρα αναδιάθρωση. Ο συνδυασμός των δύο στοιχείων λοιπόν είναι κάτι που εξετάσαμε ακροθυγώς στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα τον κύριο Λάγκεν του ΕΛΚ έχω. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Έχω μια σύντομη ερώτηση. Σε σχέση με τις προδιαγραφές ιδίου κεφαλαίου για τις τράπεζες και τις αποφάσεις βασιλείας, συζητούμε και επιμένουμε πάντοτε ότι ε, τα κρατικά ομόλογα έχουν να κάνουν με μηδενικό κίνδυνο. Αυτό είναι ένα ζήτημα της ε, ε, σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος, διότι βλέπουμε ότι οι τράπεζες δεν έχουν ε, περιορίσει το πρόβλημα, αλλά το έχουν ενισχύσει. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, η περίπτωση που προτείνετε εσείς, η λύση που προτείνετε εσείς, θα ενισχύσουν το πρόβλημα ή θα το περιορίσουν. Απάντηση εάν δημιουργηθεί ένα μέσον διαφοροποιημένου κινδύνου, με ένα διαφοροποιημένο μείγμα δηλαδή. Το πρόβλημα αυτό της, της εξάρτηση, εξάρτησης μεταξύ της χρηματοδότησης των κρατών και των επενδύσεων των τραπεζών θα είναι πιο περιορισμένο ή και μηδενικό. Τώρα το αν σταθμίζεται ως μηδενικός ο κίνδυνος από το κρατικό χρέος έχουμε σαν απάντηση ότι χρειάζεται ένα ασφαλές πεδίο για κάθε τύπο χρέους και ξέρετε ότι αυτή η στάθμιση μηδενικού κινδύνου για τα κρατικά ομολόγα ήταν μια ε, παγκόσμια συνένεση και όχι μόνο ευρωπαϊκό εφεύρημα. Εάν όμως στην Ευρώπη έχουμε την εισαγωγή διαφορετικής στάθμισης κινδύνου για τα κράτη, τότε εισάγεται σύστημα, ε, στοιχείο αστάθειας, αποσταθεροποίησης στο σύστημα. Και άρα η σταθερότητα που με πολλές προσπάθειες και κόπους έχει, επι... έχει εξασφαλίσει αυτά τα τελευταία χρόνια θα ανατραπεί. Κύριε Λάγκεν, ναι, σωστά το λέτε ότι ήταν ε, παγκόσμια συμφωνία, εθνή συμφωνία, αλλά δεν είναι κάτι το παλιό, είναι κάτι το οποίο επευλήθη με την επικράτηση της αμερικανικής ε, φιλοσοφίας περί τα δημοσιονομικά. Και συμφωνώ ότι μπορεί να καταρρεύσει ο τραπεζικό τομέα, ε, ε, αλλά από την άλλη συμφωνούμε και ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, ανεξάρτητα από την Ευρωζώνη και ανεξάρτητα από, την, από το υψηλό χρέο των επιμέρου βιομηχανικών κρατών. Παρακαλώ, σύντομα θα συμφωνήσω ότι θα ήταν σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα όπου θα σημαίνει συνεγερμός πολύ πιο νωρίς από ό,τι μέχρι τώρα. Και άρα θα επαγρυπνούμε πολύ πιο νωρίς για το ενδεχόμενο ε, ελλείμματος για τα κράτη που θα μπορούσαν να οδηγήσει σε αποσταθεροποίησή τους. Μπορούμε βεβαίως να συζητήσουμε το τι είδους δεσμεύσεις μπορούμε να ζητήσουμε από τις τράπεζες, πόσο μεγάλα δάνεια δηλαδή, αλλά από την άλλη πρέπει να γνωρίζουμε και ποιος θα διακρατά τα κρατικά ομόλογα. Γιατί πάλι θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη αυτή και στο μέλλον να πολλούνται, να διατίθενται και αυτά θα τα διακρατούν είτε οι τράπεζες είτε ο πολίτης, είτε κάποιος άλλος επενδυτής, ασφαλιστικές εταιρείες, ε, ε, χαρτοφυλάκια και το καθεξής. Πάντως το βασικό είναι να υπάρχουν εγκαίρως οι δυνατότητες για το σήμα κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες δεν έγινε αυτό. Και το διαπιστώσαμε και κατά την ε, επεξεργασία του fiscal governance της οικονομικής διακυβέρνησης. Κυρία Μπενασίρ, πολύ σύντομα. Ναι, μια εναλλακτική για τη στάθμιση των κρατικών ε, ομολόγων στα ισοζύγια των τραπεζών ε, θα ήταν ένας κανόνας μέγιστης έκθεσης που μπορεί να εφαρμοστεί με πιο προοδευτικό τρόπο και να εισαχθεί στην Ευρωζώνη. Το πρόβλημα θα είναι μετά το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού με τις τράπεζες από άλλα μέρη του κόσμου. Τελικά όμως αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια για όλες τις μεγάλες τράπεζες. Κύριος Μπίσοπ, το HQLA, τα, το ρευστό ενεργητικό υψηλής ποιότητας των τραπεζών που μπορεί να πάρει τη μορφή των ευρωομολόγων θα μπορεί να είναι το πιο ασφαλές και ως αυτό το πιο ρευστό ενεργητικό στην Ευρωζώνη. Πέραν αυτού, εάν έχουν ε, μακροπρόθεσμης διάρκειας ε, ομόλογα στα χέρια τους οι τράπεζες, θα πρέπει ίσως να δούμε μήπως αυτά μπορούν να περάσουν σε ιδιώτες και το καθεξής. Δηλαδή θα πρέπει να αποθαρρύνουμε τις τράπεζες από αυτή την επιλογή και θα πρέπει το χρέος αυτό να μεταφερθεί στην αγορά, ασφαλιστικέ εταιρείε, συνταξιδοτικά ταμεία, όπως είπατε και εσεί απευθεία στον πολίτη. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Πρέπει κάπου να πάνε αυτά ομόλογα. Αλλά από την άλλη θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε τις τράπεζες στο μέσο δυνατό βαθμό με υψηλής ποιότητας ενεργητικό, ρευστότητα μέσω του Eurobond, του Eurobond, ευρωομολόγου. Ευχαριστώ. Η κυρία Ποδηματά έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τα μέλη της ομάδας συμπρογνωμόνων. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την ερώτηση του συναδέλφου Φίλιπ Λάμπερτς και είναι η εξής ερώτηση. Εσείς προτείνατε να προχωρήσουμε μια διακυβερνητική συμφωνία για την έγκριση του πακέτου αυτού. Η πρόταση αυτή έχει σαν στόχο να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία ως εναλλακτική σε μια τροποποίηση της συνθήκης που είναι πιο περίπλοκη και χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο. Δεύτερον, και σχετικό με το δικό σας συμπέρασμα στην έκθεση, που διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι οι χώρες του προγράμματος, εάν εξαιρεθούν από το Ταμείο Αποπληρωμής, μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο σοβαρά προβλήματα εάν κληθούν να αυτοχρηματοδοτηθούν από τις αγορές, να στήσουν χρηματοδότηση από τις αγορές. Και λέτε, χωρίς βέβαια αυτό να είναι στο πνεύμα της αρχικής εκθέσεως και το αναφέρω ως μια θετική εξέλιξη, λέτε λοιπόν και προτείνετε οι χώρες προγράμματος ε, να ενταχθούν ή ότι πρέπει να ενταχθούν, άπαξ και από το πρόγραμμά τους, στο σύστημα του Ταμείου Αποπληρωμή. Αυτό είναι πολύ καλό βέβαια για όλε τι χώρε του προγράμματο. Η Ιρλανδία έχει βγει από το πρόγραμμα, η Πορτογαλία ετοιμάζεται και ξέρετε ότι υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου που θα κριθεί με στου επόμενου μήνε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω υπό το φως αυτής της συζήτησης και με τις αναλύσεις σας και τα διάφορα μέσα εργαλεία που μας προτείνετε μαζί με τους νομικούς περιορισμούς που συνεπιφέρουν τι πιστεύετε ότι μπορεί και πρέπει να γίνει βράχη και μέσο πρόθεσμα ώστε να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του χρέους αυτών των κρατών και να διευκολυνθούν οι χώρες αυτές στην ε, διασφάλιση πρόσβαση στην αγορά και επίσης προς την αιρεσιμότητα της προϋποθέσεις. Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται την ανάγκη να είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις στην περίπτωση του Συμφώνου για την Ευρωπληρωμή του Χρέους. Έχουμε ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο για τη δημοσιονομική εποπτεία στην Ευρωζώνη, με την νέα οικονομική διακυβέρνηση, με το Fiscal Compact. Διερωτώ με λοιπόν, το πλαίσιο αυτό δεν αρκεί για να εξασφαλίσει ότι θα αντιμετωπιστεί ένας οποιοδήποτε επιπλέον κίνδυνος. Γιατί νομίζω ότι η Ευρωζώνη πάντα προχωράει με το σύστημα του μπαστούνιου και του καρότου, των κυρώσεων δηλαδή και των κινήτρων, αλλά τώρα πιο, πολλά, πιο πολλές κυρώσεις βλέπουμε παρά καρότα, κίνητρα. Απάντηση. Ναι, το κίνητρο θα ήταν, το καρότο δηλαδή, θα ήταν η κοινή έκδοση και η δυνατότητα να υποφεληθούν κυρίως από αυτό οι χώρες με το υψηλότερο χρέος. Η άλλη βέβαια όψη είναι ότι ενέχει και τον κίνδυνο σε ένα τέτοιο εγχείρημα είναι πολύ κίνδυνοι. Κάτι που δεν συζητήσαμε αλλά το έχουμε αναφέρει στην έκθεση είναι ότι τα εθνικά σύνορα και κυρίως τα εθνικά συντάγματα ορίζουν ε, περιορισμούς, ε, ε, ορίζουν όρια ως προς το τι μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και εκεί ακριβώς είναι ο κίνδυνος. Ε, αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες λοιπόν θέλουν να περιορίσουν αυτό το στόχο και να περιορίσουν τον κίνδυνο. Και με ρωτάτε αν δεν έχουμε αρκετέ διασφαλιστικέ δικλείδε ε, ήδη. Η απάντηση εκ μέρου τη ομάδα μα είναι ότι πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό υπόθηκε νωρίτερα ότι θα πρέπει να αντληθεί η σχετική εμπειρία από το ισχύον πλαίσιο διακυβέρνησης που θέσπισε το Κοινοβούλιο σας και η Επιτροπή σας τα τελευταία χρόνια. Από εκεί θα δούμε αν αρκεί, έχοντας συλλέξει την εμπειρία για δε την ε, ταχύτητα εφαρμογής. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα, η διακυβερνητική φαίνεται να είναι η μόνη λύση. Αλλά ξέρουμε ότι και αυτό θα είναι δύσκολο. Και επίσης για τις χώρες που έχουν προσαρμοστεί μέσα από ένα σύστημα Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίηση και Διεθνού Πνευματικού Ταμείου. Και αν βγουν από το πρόγραμμα, μπορούν να μπουν στο σύμφωνο απόσβεση χρέου. Ε, για οποιαδήποτε χώρα δεν υπάρχει σοβαρό, σοβαρή αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του χρέους, δηλαδή για οποιαδήποτε χώρα θεωρείται ότι μπορεί και με το ταμείο αυτό, με μια κάποια ε, υποστήριξη για την ρευστότητά της ε, μπορεί να λειτουργήσει, αλλά πάλι υπάρχουν οι αμφιβολίες. Δηλαδή δεν θα ήταν συνετό να ενταχθούν χώρες όπου μπορεί ακόμη να χρειαστούν κάποια στιγμή αναδιάρθρωση. Δεν θα πρέπει να μπουν στο Ταμείο. Διότι θα απαιτείται ένα υπερβολικά υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα για τις χώρες αυτές. Με την ολοκλήρωση όμω του προγράμματο οικονομική προσαρμογή, κανονικά θα πρέπει να μπορούν οι χώρε να μπαίνουν στο ταμείο αποπληρωμές. Για δε το συγκεκριμένο ερώτημα που συζητήσαμε στην ομάδα, τι γίνεται με το υπολοιπόμενο χρέο από το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίηση, Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί είναι ήδη η αρμοδιότητα και η ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και η ερώτηση και η απάντηση ήταν πολύ μακροσκελής, δεν έχω άλλο χρόνο και θα περάσω στην επόμενη ερώτηση της κυρίας Μπέρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της ομάδας εργασίας, ευχαριστώ για αυτή τη μελέτη, την περιμέναμε πώς και πώς, με μεγάλη ανυπομονησία, περιέργεια, μας άνοιξε την όρεξη θα έλεγα. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτη, η δεύτερη φράση των συμπερασμάτων όπου δίνεται την αναφορά ότι ουσιαστικά δεν έχουμε αρκετά πειραματιστή... δεν έχουμε αρκετή εμπειρία όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης για να μπορούμε να αποφασίσουμε περισσότερο όσον αφορά τις ανάγκες που υπάρχουν για το μηχανισμό αμοιβεοποίησης ε, με μπερδεύει. Διότι αν πιστέψω τα στοιχεία, τα αριθμητικά που διάβασα, που δημοσιεύτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον Μπρούγκελ για τις τάσεις όσον αφορά την ανεργία και τον ε, σταθερό χαρακτήρα που υπάρχει, ε, σταθερότητα και εντός της ενώσεως αλλά κυρίω στην Ευρωζώνη, στα επίπεδα, βλέπουμε ποια είναι η τάση. Η τάση δεν έχει αντιστραφεί. Άρα θα πρέπει να κάνουν περισσότερα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα καρότου ή άλλη μεθόδου που να χρησιμοποιηθεί για να εξισορροπήσουμε τα δεδομένα και να είμαστε σίγουροι ότι οι συνθήκες αλληλεγγύης ε, εφαρμόζονται προς εξυπηρέτηση μιας στατικής ανάκαμψης. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, από ό,τι κατάλαβα, αναφέρεστε στις γνωστές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, δηλαδή τα όρια που θέτουν οι συνθήκες. Και στη συζήτηση, αυτό, ε, στη συζήτηση αυτή τα όρια τη συνθήκη ήταν αποφασιστική σημασία και στο Ευρωκοινοβούλιο αποδείχτηκε ότι ακόμα και εντό των συνθήκων δεν θα πρέπει να προσφεύγουμε συνεχώ τη διακυβερνητική μέθοδο. Βλέπω έναν κίνδυνο σε μια λύση που εδράζεται επί κυβερνητικών εγγύσεων. Είναι ο ίδιο κίνδυνο με αυτόν που καταγγέλουμε όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση. Δηλαδή, ποιο είναι ο κίνδυνο. Ουσιαστικά να αντιμετωπίζουμε αντίφαση προτινομένων διατάξεων. Προτείνουμε ένα μηχανισμό για να εξισορροπήσουμε τις ε, ευκαιρίες εντός της Ευρωζώνης, να καλύψουμε τις ανισορροπίες κλπ. Ξέρετε τέλος πάντων, την έχουμε δει την ταινία. Όταν εισάγουμε αυτή τη διακυβερνητική εγγύηση, επανεισάγουμε το τρόπος τον χαρακτήρα αυτών των ερωτηματικών του μηχανισμού. Μήπως καλύτερα θα ήταν να μας βοηθήσετε να κάνουμε μεταρρύθμιση των συνθήκων που χρειαζόμαστε και εν πάση περιπτώσει εκείνοι που είναι αντίθετοι στην μεταρρύθμιση ε, ας ε, απευθύνουν εκκλησιαλού. αλλού. Δηλαδή, έχουμε προοπτική μεταρρύθμιση των συνθήκων, αλλά μας αποθαρρύνουν. Λένε ότι αυτή ε, πραγματικά δεν υπάρχει θέληση να γίνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι που δεν τη θέλουν, μας λένε απ' την άλλη ότι θέλουν μεταρρύθμιση των συνθήκων. Μία λένε το ένα, μία λένε το άλλο. Λοιπόν, αν το πούμε θέλετε τη μεταρρύθμιση των συνθηκών, που τη θέλετε, σαν αντάλλαγμα εμεί θέλουμε εκείνο. Και έτσι διοργανώνουμε ένα deal και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο παρά να λέμε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Τρίτον, γιατί υποβόσκει στη συζήτηση. Μιλήσαμε για ανισορροπίες της Ευρωζώνης κλπ. Και, και υπάρχει και άλλος μηχανισμός που καλύπτει τις ίδιες ανησυχίες. ελάχιστο επιδόματος ανεργίας. Είναι εικονοκλαστική ίσως η προσέγγιση μου που ξεπερνά την εντολή που σας δόθηκε. Λέω όμως, αφού τελειώσατε το έργο σας, μήπως μας πείτε κοιτάξτε από την άλλη πλευρά θα είναι πιο εύκολα. Ιδού, μας μένει ένα λεπτό για να απαντήσετε. Σε ποιον να δώσω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Να ξεκινήσω με το δεύτερο ερώτημα. Ίσως είναι και το ευκολότερο να απαντηθεί. Έχουμε κάνει διάκριση μεταξύ του παρόντος πλαισίου των συνθήκων, αν υπάρχει κάποια λύση εντός αυτού του πλαισίου, του παρόντος, θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιήσουμε ένα άρθρο των συνθήκων και να το συνδυάσουμε με διακυβερνητική συμφωνία. Στη διακυβερνητική συμφωνία Συμφωνώ πλήρως μαζί σας ότι είναι κίνδυνος αυτός για την Ένωση αν υπονομεύσουμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και δημιουργήσουμε παράλληλη δομή διακυβέρνησης με όλα τα προβλήματα ελέγχου, έλλειψης ελέγχου που συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Και αλλάζοντας και την κατανομή των εξουσιών. Συμφωνώ απόλυτα και περιγράψαμε το εφικτό και τι απαιτεί αλλαγή των συνθήκων να αλλάξουν οι παραδόσεις και στοιχεία όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλα αυτά απαιτούν αλλαγή των συνθήκων. Θέλαμε να περιγράψουμε δύο διαφορετικά ενδεχόμενα, αλλά δεν ε, προτείναμε, δεν ήμασταν κατά της αλλαγής συνθήκης. Τρίτον, Ίσως είναι το ερώτημα αυτό συνδυάζεται με το πρώτο ερώτημα. Βεβαίως έχουμε τεράστια προβλήματα έλλειψης, ανάπτυξης, μικρών επενδύσεων, χαμηλών επενδύσεων. Αν δείτε τα στοιχεία για τις επενδύσεις τους τελευταίους μήνες και τα προβλήματα της ανεργίας, έχουμε πρόβλημα, ναι. Βέβαια, συμπληρωματικοί μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου θα βοηθούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Να έχουμε όμως υπόψη επίσης ότι θα πρέπει να πληρώσουν τα χρέη τους οι χώρες. Μπορούν να το κάνουν αυτό ανάλογα με τα spreads που υπάρχουν βέβαια μεταξύ κρατικών ομολόγων. Μπορούμε να βοηθήσουμε να μειωθεί το άχθος αλλά δεν απαλλάσσεται το βάρος που υπέχουν τα κράτη ε, και το βάρος αυτό ε, δεν διανέμεται ισότιμα. Ο κύριος Μπίσοπ ίσως θέλει να πει κάτι. Δεν προβλεπόσασταν. Είχαμε εξαντλήσει το χρόνο. Ο κύριος Μπίσοπ, σύντομα. Εγώ αναφέρθηκα στην ανάγκη διακυβερνητικής συμφωνίας. Ανέφερα τα επιχειρήματά μου, δεν θα τα επαναλάβω. Δεν ήθελα να ακούσω άλλες ερωτήσεις καλύτερα. Ο κύριος Σμιτ. Ε, η κυρία Τάισεν ε, και εγώ ε, υποβάλαμε ερωτήσεις εκτός Ευρωζώνης. Γιατί να σκάμε και πολύ. Εάν θέλετε και άλλοι να προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη, αυτό είναι θέμα ύψης της σημασίας. διάβασα τα συμπεράσματα, σας ακούω εδώ και δύο ώρες. Μα τι θέλετε επιτέλους γιατί αν ε, διαβάσετε τα συμπεράσματα, αυτό κάνει ο δημοσιογράφος, γιατί αυτό είναι και το σπουδαιότερο, αναφέρετε ότι δεν ξέρετε αν αυτό είναι καλό ή κακό. Θέλετε περισσότερα στοιχεία, αυτό μας λέτε σε τελευταία ανάλυση. Δηλαδή πόσο πραγματικά έχετε δεσμευτεί και εδώ αποτείνομαι στο φιλανδό μου φίλο γιατί ξέρετε ότι στη Βαλτική αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε σχέση με τα νομίσματα. Είσαστε πραγματικά, δηλαδή ποια είναι η δέσμευσή σας εμείς ε, περιγράψαμε τα πιθανά ευεργετήματα και στα δύο σχέδια, αλλά αναφερθήκαμε και στη μεγάλη δέσμευση που χρειάζεται για να κινηθούμε προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Δεν θέλουμε να υποτιμήσετε τους ε, κινδύνους αν συσταθεί ένα τέτοιο σύστημα, το, ένα, το πρώτο ή το δεύτερο. Σε αυτή την περίπτωση δεσμεύεστε για δεκαετίες και εδώ γίνονται εικασίες για διάφορα σενάρια. Μπορεί να δημιουργηθεί και επιπρόσθετο άχθος και ανισορροπίες, αστάθειες και γι' αυτό θα πρέπει να μελετηθεί εις βάθος. Μα δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο εδώ. Εάν ε, συλλέξουμε στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αυτής της διακυβέρνησης, τότε θα αποφασίσουμε για οποιοδήποτε σχέδιο έκδοσης. Εάν διαβάσετε όμως ε, το, τον κατάλογο συμπερασμάτων που αφορά αρκετές σελίδες, τότε ε, καλύπτουμε κάθε πτυχή. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν έχουμε ε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε την έκθεση ούτε τα συμπεράσματα πριν από τη συζήτηση και αυτό καθιστά τα πράγματα δύσκολα. Ευχαριστώ όμως την Πρόεδρο και τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων καθώς και τα μέλη της Επιτροπής. Η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και η Επιτροπή θα αποφασίσει Δηλαδή είναι στη διακριτική ευχέρεια να μας πει ποια συνέχεια θα δοθεί σε αυτή την έκθεση. Θα το δούμε κατά την επόμενη φοιτεία. Εγώ απλούστατα ήθελα να πω αυτό που μου έκανε εντύπωση. Είπατε εσείς οι εμπειρογνώμονες ότι χρειάζεται μεγάλη εμπιστοσύνη σε σχέση με τη δέσμευση των κυβερνήσεων μακροχρόνια. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μιλάτε για μακροχρόνια δέσμευση των κυβερνήσεων, μα είναι κάπως δύσκολο, διότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν κάθε 4-5 χρόνια. Άρα ε, τι σημαίνει μακροχρόνια για σας. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω εν είδη συμπεράσματος είναι ότι κατανοήσαμε για άλλη μία φορά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στη δημοσιονομική πειθαρχία εάν θέλουμε να μειώσουμε το καλπάζον χρέος που πραγματικά είναι καλπάζον σε ορισμένα κράτη. Έχουμε μέσα το 2 το 6-pack που έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά όλα αυτά δεν λειτουργήσαν. Αν ε, ρωτήσετε λοιπόν τις ε, κυβερνήσεις, αν ζητάτε από τις κυβερνήσεις δεσμεύσεις ε, για τις κυβερνήσεις που ζουν πάνω από τα μέσα που διαθέτουν, τότε αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ίσως θα πρέπει να εξεύρουμε μια άλλη δυνατότητα να βγούμε από το στόμα του λύκου. Θα πρέπει να υπάρξει επιμερισμός κινδύνων και νομίζω ότι υπάρχει αρκετή αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Θα δούμε τι θα κάνουν το επόμενο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ε, παρεμβήκατε και για την ε, εργασία σας. καλή επιστροφή. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που ήθελα να παρέμβουν, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο στη διάθεσή μας. Και τώρα περνάμε στο σημείο 3, που είναι οι ανακοινώσεις ε, της Προέδρου. Και επειδή όλα έχουν ε, ετοιμαστεί στα αγγλικά, θα σας τα διαβάσω αγγλικά, τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Σας είπα, δεν έχω οξφορδιανή προφορά ή προφορά Cambridge, γι' αυτό ζητώ κατανόηση. Θα ήθελα να πληροφορήσω όλα τα μέλη, ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι η φωτογραφία θα γίνει 7 Απριλίου στις 5 παρατέταρτο για να έχουμε την ομαδική φωτογραφία των ε, μελών της ΕΚΟΝ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα υπόλοιπα είναι εξίσου σημαντικά. Τι γίνεται με τους τριμερείς διαλόγους. Το, το Κοινοβούλιο σε σχέση το, με το MR έλαβε αποφάσεις για τις ε, καταχρήσεις στην αγορά το Σεπτέμβριο και την οδηγία ε, στις, καταχρήσεων ε, στις αγορές στις 4 Φεβρουαρίου και φτάσαμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο πριν από την επαλήθευση των κειμένων. Τώρα η νομική υπηρεσία και οι γλωσσομαθείς νομικοί ε, υπέβαλαν το κείμενο και έχετε το διορθωτικό της Ολομέλειας της Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ σύμφωνα με τον κανονισμό. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, το διορθωτικό θα υποβληθεί στην πρώτη σύνοδο της Ολομέλειας της Βρυξέλλες και θα εγκριθεί εκτός και αν ζητηθεί κάτι διαφορετικό από 40 μέλη ή μία ε, πολιτική ομάδα. Το κατανοήσατε ωραία. Τώρα τα υπόλοιπα. Ε, οδηγία λογαριασμών ε, πληρωμών. Φτάσαμε σε συμφωνία με βάση το τριμερή διάλογο στις 20 Μαρτίου. Τα πρώτα στοιχεία ε, επιφέρουν την ευθύνη στα κράτη-μέλη να ορίσουν ένα σύστημα για την ε, ε, πρόσβαση ενός λογαριασμού πληρωμών για τους καταναλωτές για να υπάρχει διαφάνεια και συγκρισιμότητα για αυτούς τους λογαριασμούς με βάση τις καταβολές που θα γίνουν έτσι ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν οι λογαριασμούς, οι καταναλωτές, πέρα από τα σύνορα, η Κορεπέρ, θα εγκρίνει το κείμενο στις 4 ε, Απριλίου και θα γίνει επαναδιαβούλευση της Επιτροπής ΕΚΟΝ σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού, έτσι ώστε να εγκριθεί στη δεύτερη σύνοδο του Απριλίου. Εντάξει. Τώρα, στο σημείο 4, έχουμε τους κανόνες για την ε, εξήγηση πιστοτικών Με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. Πάντα όλα αλλάζουν. Πρόκειται για νέα ε, διαβούλευση με την Επιτροπή Δυνάμει του άρθρου 70 του Κανονισμού. Η κυρία Έλσα Φερέιρα ε, είναι η συγγήτρια, δεν με ακούει. Η Σκιώδης είναι η κυρία Κόριν Βόρτμαν Κόλ, ε, Τόμας Χέντελ, ε, Γκουλάρ και ξέρετε ότι επήλθε συμφωνία ως προς το SRM στις 20 Μαρτίου μετά από 16 ώρες διαπραγμάτευσης και θεωρήθηκε ότι το εκτελεστικό συμβούλιο θα ασχοληθεί με όλες τις πτυχές του μηχανισμού εξυγίανσης και το, η Ολομέλεια θα αποφανθεί για τη χρήση του μηχανισμού. Χρειάζεται αυτή η διαδικασία λήψη αποφάσεων έτσι ώστε ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης να αποφασιστεί. Το Συμβούλιο θα συμμετέχει μετά από αίτημα της Επιτροπής για να ορίσει τα κριτήρια δημοσίου συμφέροντος για να μιλήσουμε για διαφορετική χρήση του Ταμείου. Συμφωνήθηκε ότι η δυνατότητα δανειοδότησης θα προωθηθεί και η περίοδος αμοιβεοποίησης θα μειωθεί από 10, από 10 σε 8 χρόνια. Αρχίζοντας με 40% το πρώτο έτος και 20% το επόμενο. Ο τριμερής αυτός διάλογος ε, ακολουθήθηκε ε, από έναν άλλον στις 24 Μαρτίου για τα μείζωνα πολιτικά ζητήματα και ε, οριστικοποιήθηκε στις 25 ε, Μαρτίου. Ελήφθη μια επιστολή από την Κορεπέρ στις 28 Μαρτίου και διανμήθηκε στα μέλη της ΕΚΟΝ. Θα γίνει νέα διαβούλευση σε σχέση με το κείμενο του Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην Ολομέλεια ε, στις 9 Απριλίου και θα ψηφιστεί στη δεύτερη Ολομέλεια του Στρασβούργου. με όλους τους αρμόδιους φορείς. Το κείμενο που θα ψηφιστεί ε, δεν είναι ε, ένα τελικό κείμενο και θα πρέπει να αναθεωρηθεί από νομομαθείς από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Μαΐου, όπου θα γίνει νέα διαβούλευση των ε, μελών με βάση τη γραπτή διαδικασία για το διορθωτικό. Το διορθωτικό θα ανακοινωθεί στη δεύτερη ολομέλεια του ε, Ιουλίου και θα εγκριθεί εκτός και αν υπάρξουν αντιρρήσεις μέσα σε 24 ώρες. Το τελικό κείμενο του Συμβουλίου και η υπογραφή του κανονισμού θα γίνει τον Ιούλιο ή το Σεπτέμβριο και το κείμενο θα δημοσιευθεί στην ε, επίσημη εφημερίδα μετά την υπογραφή του. Τώρα θα ήθελα, δυνάμει του άρθρου 70, να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας. Συμφωνείτε? Εάν θα πρέπει να ψηφίσουμε, δεν θέλει να παρέμβει κάποιος? Ε, λοιπόν, ψηφίζουμε διανατάσεως. Νομίζω ότι υπάρχει ε, πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία. Εντάξει. Ο η εισηγήτρια θέλει το λόγο, η κυρία Φερέιρα θέλει κάτι. Ναι, έχετε, έχετε το λόγο διαδικαστικό. Κύριε Λάγκεν, το περιεχόμενο αυτού που πακέτου με ενδιαφέρει το είναι το γεγονός ότι η στάθμιση των ε, πληρωμών ε, με βάση τον κίνδυνο θα πρέπει να ενταχθεί μέσα σε ένα κανονισμό του Συμβουλίου. Να τα επαναλάβετε παρακαλώ. Η ερώτησή σας ήταν, η ερώτησή μου ήταν εάν οι εισφορές των επιμέρους τραπεζών, μικρών μεγάλων, με βάση τη στάθμιση του κινδύνου, μπορεί να ενταχθεί σε ένα ε, κανονισμό του Συμβουλίου και να ρυθμιστεί στις λεπτομέρειες, στις τεχνικές λεπτομέρειες. Did you get it? Κύριος Γκίγκολτ, εντάξει, το καταλάβατε. Όχι, εμένα, εμένα να λέτε. Ε, τουλάχιστον, τουλάχιστον να αισθανόμαστε όταν μιλάμε και οι δύο γερμανικά. Ε, ναι, αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει, αλλά έχουμε μαζί από κοινού διαβουλευθεί. Και έχουμε λάβει από την Επιτροπή την απάντηση ότι για την Επιτροπή ε, για την οδηγία εκαθάρισης θα πρέπει να υπάρχουν κατεξουδότηση πράξεις ώστε να προβλέπεται και για το Κοινοβούλιο η δυνατότητα να αμφισβητήσει τις αποφάσεις αυτού του κανονισμού. Το πρόβλημα θα είναι ότι ο κανονισμός θα αποφασίζει, ο κανονισμός του Συμβουλίου, να μοιράζει 55 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι το οποίο εμείς είχαμε πει ότι δεν είναι σκόπιμο για ένα κανονισμό του Συμβουλίου. Η δυνατότητα που έχουμε είναι με το ένα πακέτο, με τις καταξιδότητες πράξεις, να επανακτούμε τον έλεγχο των αποφάσεων στα τεχνικά στοιχεία. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα στην προσεχή θητεία, διότι τελικά οι μικρές τράπεζες θα επιδοτούν τις μεγάλες και τις τράπεζες επενδύσεων. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι σύστημα σταθερότητα. Η πρόεδρο. Ναι, αλλά μάλλον δεν θα γίνει αυτό τον Ιούλιο. Δύο μήνε μα μένουν μόνο. Το Σεπτέμβριο πρέπει να πάει. Και άρα εμεί δεν έχουμε τίποτα να πούμε σε αυτή την υπόθεση. Κατεξουδότηση πράξη είναι μια παράξενη ιστορία, παράδοξη και για άλλε επιτροπέ. Και πρέπει εμεί να βεβαιούμαστε ότι η απόφαση με της πράξης έρχεται μόνο Σεπτέμβριο και έχει πιο νωρί. Ναι, αλλά έχει δώσει υποσχέσει η Επιτροπή και βεβαιώσεις με τελευταία διάσκεψη των συντονιστών. Καλά, έστω εγώ δεν είμαι μέλος των συντονιστών και δεν γνωρίζω. Κύριος Λάγκεν, αντίθετα από τον κύριο Γκίγκολτ, εγώ θεωρώ ότι η απόφαση συμβουλίου, το κανονισμό συμβουλίου δηλαδή, είναι μια λύση καλή γιατί θα μας κερδίσει και κανένα δύο μήνες και επίσης διότι το συμβούλιο θα βρει μια ε, λύση ικανοποιητική για μας, μια ορθολογική λύση στάθμισης του κινδύνου. Καλώς λέει η Πρόεδρος. Εν πάση πτώση είπατε ότι συμφωνείτε, έχετε ψηφίσει και ως εκ τούτου τα πράγματα τα αφήνουμε να πάρουν την πορεία του. Με την ελπίδα ότι το Κοινοβούλιο θα αρκετεί ο χρόνο στη θεσή του όταν έρθει να δει αυτές τις πράξη, να μην χάσει τον έλεγχο των όσων έχουν αποφασιστεί στο Συμβούλιο και στον τριμερή διάλογο, γιατί πάντα παραμένει αυτό ο κίνδυνο. Κυρία Φόρτ. Πόσο μιλάμε γι' αυτά, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που είπατε ότι τώρα και τα τρία νομοθετήματα θα ψηφιστούν από κοινού. DGS, RAD ε, και SRM και προφανώς επ' αυτών των θεμάτων το πώς κάθε θεσμικό όργανο θα συμβάλλει αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για Λάγκεν το προηγούμενο που δημιουργήθηκε στην ενιαία αγορά δηλαδή η καταξιοδότηση πράξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να γίνεται σεβαστό και σημειώστε κυρία Πρόεδρε για τα πρακτικά ότι θα ήταν καλό να συμφωνηθεί στον κατάλογό σας το συμπεφωνημένο διακυβερνητική συμφωνία με άλλα λόγια που μεταξύ άλλων καλύπτει με και τα μη, την αντιμετώπιση των μη συμμετεχόντων κρατών μελών. Θα σημειωθεί αυτό που προτείνατε. κυρία Φερέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη διότι δεν άκουσα την ερμηνεία που εδόθη τη ερώτησης του συναδέλφου. Ε, τον ευχαριστώ διότι απάντησε. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω για την στενή συνεργασία και τη σοβαρή συνεργασία από όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα από τους σκιώδεις. Έτσι, το Κοινοβούλιο είχε ενιαία θέση στις διαπραγματεύσεις και βελτιώθηκε το κείμενο του Συμβουλίου. Θα ήθελα να τονίσω ότι μαζί με αυτές τις κατεξιοδότηση πράξεις θα πρέπει να ζητήσουμε από το επόμενο Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγης τη διαδικασία ε, της διακυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών. Ζητήθηκε αιτήσια, ε, συγγνώμη, μηνιαία έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα ισχύσει άμεσα και από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα έχουμε μηνιαίες συνοδευτικές εκθέσεις, έτσι ώστε το Ταμείο να λάβει σάρκα και ωστά και να μπορέσει να λειτουργήσει την 1η Πρώτου 17. Η όλη διαδικασία του Ταμείου Εξυγίανσης θα ήθελα λοιπόν η επόμενη ΕΚΟΝ να παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε ε, να υπάρξει σωστή επικύρωση. Και περιμένουμε και μία δήλωση του Συμβουλίου, αυτό συμφωνήθηκε, δεν φαίνεται στα πρακτικά, αλλά έχει συμφωνηθεί ότι θα προβεί σε μία δήλωση για την επικύρωση αυτή τέλος θα ήθελα να πω ότι είτε στα άρθρα είτε στην αιτιολογική σκέψη το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να οριστεί μία ε, γραμμή πίστοσης από την αρχή της λειτουργίας ε, του Ταμείου. Αυτό είναι και χρέος της επόμενης έκον, να επιμείνει δηλαδή αυτό δηλαδή που, για το οποίο λάβαμε μια πολιτική υπόσχεση να υλοποιηθεί, διότι αυτή η γραμμή του προϋπολογισμού είναι πολύ ε, σημαντική για το Κοινοβούλιο με βάση την αγαστή συνεργασία η οποία ε, προηγήθηκε. Ευχαριστώ κυρία Συγήτρια. Δεν μπορώ παρά να σας πω ότι δεν μπορούμε παρά να ελπίσουμε ότι οι κληρονόμοι μας στην επόμενη διάσκεψη θα είναι εξίσου ε, καλοί και θα επαγρυπνήσουν όπως και εμείς για το θέμα αυτό. Η κυρία Βόλτμαν Κόλ, ζητώ συγγνώμη. Ε, ένα λεπτό υπομονή για το σημαντικότατο θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελίζα και τους ε, συναδέλφους. Ήμασταν πραγματική ομάδα και χάρη σε αυτό πετύχαμε το ιστορικό αυτό αποτέλεσμα και διεκπαιρεώσαμε αυτή την ε, Τραπεζική Ένωση πριν τι εκλογέ. Ευχαριστώ του συναδέλφου. Περάσαμε μερόνυχτα μαζί σε τριμερεί διαλόγου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη γραμματεία τη Επιτροπή ΕΚΟΝ, την Κλέρ, και του βοηθού μα που έκαναν αξιοσημείωτη δουλειά στου τεχνικού τριμερεί διαλόγου, διότι έπρεπε να διευθετηθούν πολλά τεχνική φύση ζητήματα και χάρη στην υποστήριξή του καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία και είναι ενδεδειγμένο να του ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ που διορθώσατε κάτι που λησμόνησα. Το είχα υπόψη μου. Ναι, όλο το προσωπικό έκανε μια υπέροχη δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σας πω ότι η καλύτερη απόδειξη που είδα όσον αφορά τη σημασία που έχει το Κοινοβούλιο είναι ότι μπορέσετε τηλεφωνήσατε στις 4.30 το πρωί στον κύριο Σόιμπλε για να συμφωνήσει επιτέλους. Δεν ξέρω αν αληθεύει, αυτό διάβασα. Και αν έτσι έχουν τα πράγματα, σίγουρα ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Κυρία Λούλινγκ, ε, εφόσον προχωρούμε τώρα και πάμε σε συζήτηση θα ήθελα να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ευχαριστώ το προσωπικό. Ήταν πραγματικά ευρωπαϊκή εμπειρία. Αισθάνθηκα ότι περνάω μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ήμουν μόνος άντρας, στον οποίο το επετράπη να σημαντικά ζητήματα και με αντιμετώπισαν καλά. Συνήθως με αντιμετώπισαν καλά, με καλομεταχειρίστηκαν. Πέρα από αυτό, επί της ουσίας, Νομίζω ότι ήταν σημαντική η κίνηση αυτή και έδωσε προστιθέμενη αξία το Κοινοβούλιο. Διότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που ήθελε να μας προσφέρει το Συμβούλιο. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Ε, υπήρξαν σημαντικά επιτεύγματα. Δεν γνωρίζω ποιον εκάλεσαν. Σίγουρα ο κύριος Σόιμπλε εκλήθη. Δεν λάβαμε δεν ξέρω αν υπήρξε ο κ. Μοσκοβίτσα, ήταν και άλλοι όμως, ίσως η Κορίνα το γνωρίζει. Δείχνει όμως και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου. Και είναι η μέθοδος λήψεως αποφάσεων, όπου είναι πολύ αμφισβητήσιμη. Καλούνται κάποιες χώρες, δεν καλούνται άλλες, δεν υπάρχουν κριτήρια. Δείχνει τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Δεύτερον, που θα ήθελα να θίξω, είναι το εξής. Η διακυβερνητική συμφωνία, η διακυβερνητική συμφωνία, λέγω, είναι πρόβλημα. Διότι για πρώτη φορά έχουμε δεχτεί ότι στη διαδικασία και στη συναπόφαση στη η διακυβερνητική συνθήκη θα πάρει στοιχεία από τη συναπόφαση σε διακυβερνητικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να αλλάξουν αυτά στο μέλλον. Έχουν βγει από αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε στη συναπόφαση. Είναι ένα θέμα αρχής και θα πρέπει να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Κατά πόσο θα προσφύγουμε κατά της διαδικασίας αυτής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι ίσως δημιουργηθεί προηγούμενο στο μέλλον. Ό,τι δεν αρέσει στο Συμβούλιο και ό,τι το δυσκολεύει να το συμφωνήσει μαζί μας το θέτει σε ε, διακυβερνητικό πλαίσιο μαζί με τη συναπόφαση. Σύμφωνα με τις νομικές υπηρεσίες και των τρία θεσμικών οργάνων αυτό θα μπορούσε να γίνει στη συναπόφαση. Όμως η πρόοδος για την Τραπεζική Ένωση είναι τόσο σημαντική που μπορούμε να την υπερψηφίσουμε, δικαιολογούμεθα. Η νομική όμως πλευρά και η δημοκρατική πτυχή είναι άκρως αμφισβητήσιμες μπορώ να πω ότι όλοι ήσασταν Τι θαυμάσει Το Συμβούλιο μετακινήθηκε κατά την άποψή μου, δεν κινήθηκε αρκετά. Λένε Γερμανά, ε, είναι μια τέχνη πολιτική, είναι καλύτερο να σταματήσουμε τώρα παρά να, να τα δώσουμε στην επόμενη θητεία. Εργαστήκαμε τόσο πολύ, νομίζω ότι ήταν συνετό και ευφυές να σταματήσουμε εδώ ακόμα και δεν συμφωνούμε απόλυτα. Όσον αφορά το πρόβλημα αν θέλουμε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι το Συμβούλιο υπονομεύει μονίμως τις αρμοδιότητές μας ως συνομοθέτης αυτό θα το δούμε στο επόμενο Κοινοβούλιο. Και εμείς ναι. Δεν είναι ότι και εμείς δεν το κάνουμε, αλλά από διάφορα κράτη πρέπει να πω. Και εσείς προέρχεστε από ένα κράτος με το οποίο έχουμε μια σειρά προβλημάτων, πρέπει να πω κύριε Λάγκεν. Τώρα τελειώνουμε. Αυτή την πρώτη παρουσίαση, αλλά έχουμε άλλες δύο εκθέσεις, άλλα δύο σημεία που πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Έκθεση ΣΒΑΜΠ Euh, euh, Πρέπει να σας πω λοιπόν όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Σβάμπ Αγγλιστή Αναγιγνώσκουσα Είναι ο τελευταίος τιμές διάλογος για την έκθεση του κυρίου Σβάμπ Έλαβε χώρα στις 18 Μαρτίου ο διάλογος επετεύθη συμφωνία στο άρθρο 6 αποκάλυψη στοιχείων που αφορούν διαγωνισμό άρθρο 9 εθνικές αποφάσεις κεφάλαιο 4 ε, τι γίνεται με διάφορα, διάφορα πρόσθετα, πρόσθετες δαφάνες έλαβαμε επιστολή της Κορεπέρ και λέει το Συμβούλιο θα δεχόταν τη θέση του Κοινοβουλίου αν υιοθετήσει το κείμενο το Κοινοβούλιο όμως υπήρξαν κάποια λάθη στο κείμενο του Συμβουλίου σε σχέση με το συμπεφωνημένο κείμενο στις τέσσερις του κειμένου με τις τέσσερις στήλες και γι' αυτό το Συμβούλιο εξέδωσε διορθωτικό κείμενο και η επιστολή της Κορεπέρ και το διορθωτικό διενεμήθησαν σε όλου σας. Γι' αυτό η νέα διαβούλευση θα εδράζεται επί του συμπεφωνημένου κειμένου και που αντιστοιχεί στην διατύπωση της επιστολής Κορεπέρ μαζί με το διορθωτικό και αυτή η Επιτροπή ε, θα τοποθετηθεί επί του κειμένου ξανά σήμερα πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλεια που θα λάβει η χώρα στις 2 Απριλίου στο, στη δεύτερη Ολομέλεια του Απριλίου στο Στασβούργο. Και σύμφωνα με το άρθρο 30 του Σωτικού Κανονισμού αυτή η επαναδιαβούλευση υπόκειται σε ψηφοφορία. Τι θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν έχουν μείνει και πολλοί συνάδελφοι, δεν χρειάζεται νομίζω να ψηφίσουμε, ούτε και θα μπορούσαμε μάλλον. Α, πρέπει να ψηφίσουμε, μάλιστα. Καλώς, νομίζω ότι η Επιτροπή μας τον τελευταίο μήνα είχε να κάνει πολλή δουλειά και αυτό είχε και τις σχετικές επιπτώσεις προς τις ε, διαδικασίες που ακολούθησε η Επιτροπή κύριος Λάγκεν και άλλοι είχαν προτείνει την ε, ερώτηση αν χρειάζεται να πάει σε δεύτερη φάση αυτό το θέμα. Από τα αποτελέσματα βλέπω ότι έχουμε σοβαρά αποτελέσματα. Αλλά σας παρακαλώ να σημειώσετε, κυρία Πρόεδρε, ότι στο προσεχές κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές και διαδικασίες που ισχύουν στο Κοινοβούλιο αλλά και στη δική μας Επιτροπή, διότι είναι πολύ δύσκολο να χειριζόμαστε θέματα με τόση πίεση χρόνου, με τόση πίεση από το ε, Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο για να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και από το Κοινοβούλιο βεβαίως να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Πάντως πιστεύω ότι είναι, είναι καλά τα αποτελέσματα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και οδησίγητες του Συνολού που με βοήθησαν να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία. Χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Σλάνγκεν, μια γενική ερώτηση. Στο σημείο 4 βλέπω και διαβούλευση εδώ. Γιατί δεν λέγεται ότι πρέπει να γίνει και ψηφοφορία. Κανονικά η ψηφοφορία δεν ε, σημαίνει για τους αδέλφους ότι θα ψηφίσουμε κιόλα. Re Reconsultation. Επανα. Δεν, ε, δεν φέρω εγώ την ευθύνη όπως και να έχει. Μα ακριβώς αυτό εννοώ ότι όταν μας επιβάλλεται τέτοιου είδου ε, πίεση και δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις με τη σειρά τους και με την τάξη τους, να μην ξαφνιαζόμαστε και για τα αποτελέσματα. Όχι, όχι, και με τη σειρά τους και με την τάξη τους. Απλώς σήμερα συμφωνούμε ότι το αποτέλεσμα μπορεί να πάει για έγκριση από την Ολομέλεια. Είναι το μόνο το οποίο έχουμε να κάνουμε σήμερα. Δεν θα αναλάβουμε εμείς τώρα να την ευθύνη να παραπέμψουμε το θέμα αυτό ολόκληρο στο προσεχές κοινοβούλιο. Έχουμε προχωρήσει με έναν καλό τριμεριδιόλογο, έχουμε αποτελέσματα αποδεκτά και μπορούμε πλέον, να προχωρήσουμε. Ο κύριος Γκόβερς έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, μπορεί να είναι αποδεκτά τα αποτελέσματα, αλλά δεν γνωρίζει κανείς ποια είναι τα αποτελέσματα. η πρόεδρος μου, δεν ξέρω αν αυτό αρκεί. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, αλλά... Κύριε Σφαπ, εσείς τα ξέρετε τα αποτελέσματα. Και σας τα διάβασα κιόλας. Μα αν θέλετε, πολύ ευχαριστώ. Και τη Δευτέρα να ψηφίσουμε. Αλλά, μπορούμε μπορούμε, θα φροντίσει η γραμματεία να έχουμε το κείμενο και να ψηφίσουμε με άρση της χειρός, με ανάταση της χειρός τη Δευτέρα. Αλλού τους άλλους θα πρέπει οριστικά να γίνει προφορία στο Στρασβούργο. Λάγκεν. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι το πρόβλημα μόνο η μετάφραση, ότι δεν έχει κατατεθεί το κείμενο ή ότι κάποιος έχει να πάει διακοπές. Όχι, σας διάβασα. ότι υπήρξαν κάποια παροράματα στο κείμενο, μη αιτιολογημένα. Μπορεί φυσικά να συμβεί αυτό. Είμαστε σε έναν βαθμό με το ε, πλάτη στον τοίχο γιατί δεν θέλουμε να, να πέμψουμε όλα τα ζητήματα να τα αφήσουμε για το προσεχέ κοινοβούλιο. Ναι, αλλά αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να μα παίρνουν και στα σοβαρά πρέπει να τηρούμε του κανόνε αυστηρά, διαφορετικά θα μα πάρουν ποτέ στα σοβαρά. Καλώ λέει η Πρόεδρος, έχω ακόμα ένα αίτημα όμω για ε, εκ μέρου του κυρίου Χάνης Πέτερ Μάρτιν, ο οποίο δεν είναι εδώ, για τις ε, εμπορικέ στατιστικέ. Όχι, στο συγγνώμη. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με αυτή του προηγούμενου σημείου. Δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία διαφορετική διαδικασία γιατί όσοι συμμετείχαμε ε, ξέρουμε τη διαδικασία που, γιατί πρόκειται για επαναδιαβούλευση θα θέλαμε να αποστείλουμε στην Ολομέλεια μια συμφωνία μετά από εντολή αυτής της Επιτροπής. Δηλαδή προϋπήρξε εντολή και όσοι συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία έχουμε την, ε, τις ίδιες πληροφορίες. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να αναβάλουμε το όλο θέμα. Νομίζω ότι πρόκειται για την ίδια διαδικασία με την προγενέστερη. Τότε θα ε, επιτρέψτε μου να φέρω αντίρρηση στον ε, αξιότιμο συνάδελφο, γιατί με την έκθεση Φερέρα κάναμε τη σχετική εκδήλωση με την δήλωση του Προέδρου, πολλές ακροάσεις και εκθέσεις και εν τέλει να που καταλήξαμε τις αποφάσεις. Εδώ είχαμε αρκετή ενημέρωση και για τις δύο αυτές εκθέσεις δεν συμβαίνει το ίδιο. Ναι, ίσως, ίσως να το έχετε διαβάσει, να το είχατε διαβάσει, να το είχατε λάβει. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση αν θέλετε να ψηφίσουμε, θα ήταν ίσως καλύτερα. Αλλά τι αλλάζει εν τέλει. Ας μην ε, ξεκινήσουμε εδώ μια ολόκληρη διαμάχη δικαστικά. Αν θέλετε για τη Δευτέρα, ευχαριστώ να το κάνουμε τη Δευτέρα. Και σήμερα θα μπορούσαμε όμως όπως με την έκθεση Φερέρα και με την έκθεση ΣΦΑΠ. Απλώς πρέπει να ρωτήσω εάν πρόκειται να, αν δέχεται να ψηφίσει η πλειονοψηφία των μελών. Να ρωτήσω λοιπόν. Συνάδελφοι, ποιος θέλει να το ψηφίσει, να το εγκρίνει. Να δω αν υπάρχει αυτή η πλειονοψηφία ψηφοφορία. Εάν υπάρχει πλειονοψηφία. Μα έπρεπε να είναι μέσα στα έγγραφα, λέει ο κ. Λάγκεν. Μα τα λάβατε από το κορεπέρ, είναι τα έγγραφα του κορεπέρ που μας απεστάλησαν, μου το λέει η γραμματεία. Στην ημερήσια διάταξη για σήμερα έπρεπε να είναι. Από χτες, από χτες. το κείμενο του Κορεπέρ με το διορθωτικό μαζί είχε, έχει αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής μας. Ερωτώ λοιπόν πότε, μου λέτε εχθές. Τι να σας πω τώρα, αυτό θα αρχίσουμε να κάνουμε. Εφόσον μια πλειονοψηφία θέλει για την έκθεση ΣΦΑΠ, όπως και για την έκθεση Φερήρα, ήταν πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότεροι. Ο κύριος Λάγκεν κάνει καταμέτρηση των παρόντων. Κύριε Σφάπ, Πρόεδρε, νομίζω ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει φορλία, ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας εν τέλει εγκρίνει τη συμφωνία αυτή και τη λύση που βρήκαμε ε, προς το... ως προς αυτό λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να χανόμαστε μέσα σε δικαστικές συζητήσεις. Από την άλλη υπάρχουν διάφορα διαδικαστικά ζητήματα για το αν ψηφίζουμε εδώ ε, ενώ δεν προβλεπόταν στην ημερήσια διάταξη. Καταλαβαίνω τι λέει ο κύριος Γκέμπελς και ο κύριος Λάγεν. Από την άλλη αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στα συνέπεια που μπορεί να προκύψει για τη δουλειά των επόμενων μηνών ώστε να μπορέσουμε να, να λύσουμε όλα τα ζητήματα λοιπόν. Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου, ο κύριος Άνσερς το σημείωσε. Αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ ότι είναι σημαντικό το θέμα και πρέπει να μας απασχολήσει. Είπαμε Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Λούλινγκ. Χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, έτσι κλείνει η υπόθεση και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι με την έκθεση ΣΦΑΠ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος στην προσοχή σύνθεση της επιτροχής θα πρέπει να τον ενημερώσουμε όμως ότι πρέπει τα πράγματα να προχωρήσουν διαφορετικά από ό,τι μέχρι τώρα. Και πάω στην τρίτη έκθεση του Hans Peter Martin. Όπου πάλι έχουμε την επαναδιαβούλευση. Επί τη βάση του άρθρου 70 της διαδικασίας του κανονισμού μας. που και πάλι έχουμε καταλήξει σε μια λύση από τον τεμερή διάλογο. Ο Χάνς Πέτερ δεν είναι παρόν. Παρακαλώ όμως και εσείς να συμφωνήσετε δυνατά σωστής να αποσταλεί το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης στην Ολομέλεια. Το ίδιο πράγμα είναι. Ευχαριστώ πολύ αν συμφωνείτε. Σάντσες. Το θέμα όμως είναι το ίδιο και το ψηφίσαμε. Θα ήθελα να ε, ρωτήσω κατά πόσο ψηφίστηκε. Δηλαδή τι ακριβώς έχει γίνει. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο τα προηγούμενα έχουν ψηφιστεί. Ναι, και οι τρεις εκθέσεις θα ψηφιστούν οριστικά στην Ολομέλεια αλλά χρειάστηκε εδώ να ψηφίσουμε για την επαναδιαβούλευση, λέει η Πρόεδρος. Στα διάφορα υπάρχει κάτι. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 7 Απριλίου στη, από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλό βράδυ. Γεια σας.